Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto approviamo l'ordine del giorno. Ας δεχθούμε παρακαλώ την μερίσια διάταξη συνάδελφοι. I risultati del Consiglio di marzo 2000. Η Ουγγρική Προεδρία μας προτείνει λοιπόν να συζητήσουμε το θέμα της πολιτικής για το μέλλον της ΚΑΠ. Ο Σάντορ Φαζέκας Προσκαλείται λοιπόν για ανταλλαγή απόψεων αύριο στις 3 το μεσημέρι πριν από την συζήτηση για τις τροπολογίες της έκθεσης που προβλέπεται στην μερίσια διάταξη. Την έκθεση DES. Λοιπόν, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις άλλες, υπάρχει συγκεκριμένη τροποποίηση. Εντάσσουμε τη συζήτηση με την Ουγγρική Προεδρία στην αυριανή μας απογευματινή συνεδρίαση. Η σημερινή συνεδρίαση ξέρετε ότι αναμεταδίδεται από το διαδίκτυο. Δίνω αμέσως το λόγο αφού καλωσορίσω θερμά τον κύριο Ποτότσνικ, τον υπεύθυνο ε, για το περιβάλλον. Ο κύριος Γιάννης Ποτότσνικ έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο, όλο και πιο σημαντικό για την αγροτική πολιτική. Είναι χαρά μας η παρουσία του εδώ σήμερα στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρου και μπορεί να μας παρουσιάσει τις απόψεις του για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μετά το 2013 και για την ε, λήψη υπόψη των θέσεων τις οποίες η Γεωργία εκφράζει στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, ιδιαίτερα σχετικά με την αηφορία και την υποστήριξη στους γεωργούς. Θα δέσουμε αμέσως το λόγο στον Επίτροπο και αμέσως μετά θα ξεκινήσει εφόσον το επιθυμείτε και εσείς η συζήτηση. Ευχαριστώ Επίτροπε Ποτότσνικ, με χαρά σας δίνω το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, Αγαπητά μέλη, είναι χαρά μου να είμαι ανάμεσά σας. Χαίρομαι που έχουμε την δυνατότητα να σας παρουσιάσω τα θέματα τα οποία αποσχολούν το δικό μου χαρτοφυλάκιο στην δική σας επιτροπή. Ο πατέρας μου ήταν γεωργός και ξενοδόχος. And keeping the countryside around his well managed. Και αυτά που έμαθα από αυτόν όταν ήμουν νέος είναι να σέβομαι το περιβάλλον αλλά και τη σκληρή ζωή των γεωργών. We are living in a very fragile. Οι χρόνοι τους οποίους βιώνουμε, η εποχή θα έλεγα είναι μια έφραστη εποχή υπάρχει αλληλοδιασύνδεση και αλληλοεξάρτηση ανάμεσά μας πλέον και έχουμε γίνει ένα παγκόσμιο χωριό. Σύμφωνα με τα δεδομένα των Ηνωμένων Εθνών, τον 20ο αιώνα ο πληθυσμός αυξήθηκε τέσσερις φορές τετραπλασιάστηκε 40 φορές η οικονομική παραγωγή η κατανάλωση του νερού και η αλίευση 35 φορές, 60 φορές η κατανάλωση ε, ανθράκων και οι εκπομπές καυσαερίων 70 φορές. Βλέπουμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις θα φτάσουμε τα 9 δις στα μέσα του 21ου αιώνα σαν πληθυσμός και οι ε, καταναλώσεις θα αυξηθούν σε τεράστιο ποσοστό. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι προφανές που έχουμε μπροστά μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε πλέον με την ίδια λογική. Πρέπει να αλλάξουμε τους τρόπους παραγωγής, πρέπει να αλλάξουμε τους τρόπους κατανάλωσης και χρειαζόμαστε τη λεγόμενη επανάσταση της κοινή λογικής. Αυτό από αυτό θα εξαρτηθεί η ποιότητα του περιβάλλοντος, σε όλες τις μελέτες φαίνεται αυτό, παραγωγή ενέργειας, μεταφορικές δραστηριότητες και γεωργία. Στην έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος της αρμόδιας αρχής ε, η διαχείριση των γεών και η διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι δύο βασικά θέματα. Εγώ στην δική μου πολιτική εντολή έχω θα έλεγα τρεις βασικές προτεραιότητες. Λοιπόν, καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων, ε, βιοπικιλότητα και σωστή διαχείριση των πρώτων υλών. Εδώ αναφέρομαι στους φυσικούς πόρους, στο νερό, στα οικοσυστήματα, στη χρήση της γης, του εδάφους λοιπά Όλα αυτά έχουν συνέπειες για τους γεωργούς όπου οι πόροι κατέχουν ένα πολύ σημαντικό κεντρικό ε, τόπο θα έλεγα στην καθημερινή μας ζωή. Έχω αναφερθεί επανειλημμένα στη σημασία της γεωργίας για το περιβάλλον. Ο λόγος είναι απλός. Από κοινού οι γεωργοί και αυτοί που διαχειρίζονται τα δάση διαχειρίζονται τα τρία τέταρτα του συνολικού μας εδάφους. Ο τρόπος με τον οποίο το κάνουν αυτό είναι κρίσιμος για την επιβίωση του εδάφους, για την προστασία των υδάτινων πόρων, για την προστασία της βιοπικιλότητας και για την επίτευξη των περιβαλλοντικών μας στόχων. Το περιβάλλον πρέπει να μας προστατεύσει. Εφόσον θέλουμε εμείς να εφαρμόσουμε τα προγράμματά μας, έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρότατες δυσκολίες. Θα μπορούσε να συμφωνήσει κανείς ότι οι κατευθύνσεις που δεικνύονται από τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ εδώ από τη δεκαετία του 80 ήταν θετικές για το περιβάλλον, αλλά μένει πολλά ακόμα να γίνουν να σας μεταφέρω κάποια χαρακτηριστικά που θα ήθελα να έχει η ΚΑΠ στο μέλλον. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σχετικά με την ανακατανομή των άμεσων πληρωμών, με την ενίσχυση της αγροτικής ανταγωνιστικότητας και της σωστής ανάπτυξης της υπαίθρου. Η ΚΑΠ θα πρέπει επίσης να συνεισφέρει, η μελλοντική ΚΑΠ, στις ανάγκες μας για να καλύψουμε ακριβώς τις ανάγκες που έχουμε στον τομέα του περιβάλλοντος. Οι ανησυχίες αυτές είναι θα έλεγα σημαντικότατες για όλους τους πολίτες της Ένωσης. Νομίζω ότι τα χρήματα που θα επενδυθούν στην γεωργία μπορούν να τεκμηριωθούν εφόσον η μελλοντική ΚΑΠ συνεισφέρει και αυτή με τη σειρά της για να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους κλιματολογικούς στόχους που έχει θέσει. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές σήμερα για να αποφύγουμε μελλοντικά προβλήματα. Για να το πω αλλιώς, η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Αυτή πρέπει να είναι η μελλοντική ΚΑΠ λοιπόν. Πρέπει να είναι μια πράσινη ΚΑΠ φυσικά, μια οικολογική ΚΑΠ και αντί να επιβάζουμε κυρώσεις στους γεωργούς, επιβάλλουμε κυρώσεις σε αυτούς που δεν σέβονται τους κανόνες, θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο να αμείβουμε αυτούς οι οποίοι παρέχουν σωστά προϊόντα και τους οποίους η αγορά πολλές φορές δεν αμείβει ανάλογα. Οι μεταρρυθμίσεις από οικολογική θα έλεγα προοπτική περιλαμβάνονται και στην επιστολή που συνυπόγραψε ο Σιόλος η κυρία Χίντεγκαρ και εγώ οι τρεις επίτροποι. Πρώτον, λέμε ότι θα πρέπει να γίνουν πιο πράσινες οι άμεσες πλήρωμες επί τη βάση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών δράσεων, τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη στο σύνολο των εδαφών του η Δεύτερον, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανάπτυξη της υπαίθρου, ενισχύοντας τη σωστή εφαρμογή των ρυθμίσεων που ισχύουν επί τη βάση των προτεραιοτήτων στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 και πρέπει να υπάρξει και ένα πιο εύκολο και γραμμικό σύστημα θα έλεγα δικτών για να αξιολογούμε την πρόοδο της κατάστασης. Και τέλος ή ε, το streamlining είναι κάτι το οποίο θα ε, επιτρέψει να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις στα πλαίσια των μέτρων καταπολέμησης των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών σχετικών με τις γεωργικές δραστηριότητες. Αυτές είναι βασικά λοιπόν οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ουχή μόνο οι ειδικέ μου θέσεις. Το να γίνουν ε, οι πληρωμές του πρώτου πυλώνα πιο πράσινες θα έλεγα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί καλύπτουν ένα τεράστιο ποσοστό του κοινοτικού εδάφους. Είναι το θεμέλιο για τα ελάχιστες προϋποθέσεις που θα πρέπει να σέβονται οι γεωργοί και η Ευρώπη θα πρέπει να τους αμείβει γιατί θα λαμβάνουν μέτρα ανιχνεύσιμα τα οποία θα αποδεικνύουν ε, τον σεβασμό των κανόνων. Ε, αυτό το πρασίνισμα σε εισαγωγικά θα επιτρέψει μια καλύτερη ανάπτυξη της υπαίθρου η οποία θα συνοδεύεται από βελτιώσεις πέραν των αυστηρά νομικά προαπαιτούμενων. Ας πούμε το θέμα της βιοπικιλότητας, σαν παράδειγμα. Η επιστήμη μας λέγει ότι ζούμε μία περίοδο μαζικής εξαφάνισης ποικιλιών και οικοσυστημάτων τον προηγούμενο Μάρτιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ανέλαβαν την υποχρέωση να προωθήσουν μέτρα σεβασμού της βιοπικιλότητας και αντιμετώπισης της καταστροφής των ειδών στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 και πιθανώς αποκατάστασης εξαφανισμένων ειδών και μέσω του δικτύου Natura 2000. Ε, εδώ θα έλεγα οι χωροτάκτες των περιοχών και εκτός των προστατευομένων περιοχών, οι γεωργοί δηλαδή έχουν να παίξουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει οι χρηστές πρακτικές να εφαρμόζονται και να αμείβουμε τους γεωργούς που εξοικονομούν την χρήση του εδάφους και την χρήση των υδάτινων πόρων. Ε, συζητάω σε αυτή τη φάση με τον Επίτροπο Τσίολος ε, πώς κάποιες ε, νέες πρακτικές όπως το set aside, όπως η διαφοροποίηση των παραγωγών μπορούν να συμπεριληφθούν στα κριτήρια για τις άμεσες πληρωμές. Οι συνεχείς ε, δραστηριότητες σε βοσκοτόπια σαν παράδειγμα έχει συγκεκριμένες οικολογικές συνέπειες. Εδώ θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να δημιουργηθούν και οι βάσεις για τους λεγόμενους πράσινους διαδρόμους, έτσι ώστε τα οικοσυστήματά μας να είναι πλέον ανθεκτικά στις απειλές των κλιματολογικών συνεπειών. Έτσι θα αποτρέψουμε τη μόλυνση των υδάτινων πόρων, την διάβρωση των γεωργικών έδαφων και θα διασφαλίσουμε την ποιότητα και την παραγωγικότητα των γεών και δεν θα έχουμε ανάγκη χημικών ε, προϊόντων. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο ε, θα βοηθήσει και την καταπολέμηση των συνεπειών, την μετρίαση των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το περιβάλλον. Να προσθέσω εδώ ένα πράγμα. Οι γεωργοί και τα κράτη-μέλη συνολικά όλοι θέλουν μια πιο απλή ΚΑΠ ιδιαίτερα για το streamlining και ε, την απλούστευση των κανόνων. Συμφωνώ με τις εκκλήσεις που ακούγονται και με την ανάγκη που υπάρχει για να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην επίτευξη των δημόσιων στόχων από τη μία και τα διοικητικά προβλήματα, τα διαχειριστικά προβλήματα από την άλλη. Πολλά από τα περιβαλλοντικά θέματα στα οποία αναφέρθηκα σήμερα είναι κρίσιμα για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των γεωργών. Οι γεωργοί εξαρτώνται από σωστά και γόνιμα εδάφη, από ε, την σωστή σπορία και από τον έλεγχο των κλιματολογικών αλλαγών. Μέσω λοιπόν του πρασινίσματος σε εισαγωγικά της ΚΑΠ διασφαλίζουμε την αηφορία του γεωργικού τομέα στο σύνολό του. Πιστεύω ότι αυτό το οφείλουμε όχι μόνο στις μελλοντικέ γενναίες των μελλοντικών γεωργών, αλλά και στους σημερινούς γεωργούς και σε αυτούς φυσικά που θα ακολουθήσουν. Αγαπητά μέλη λοιπόν, η ζωή είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και προκλητική. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα μπροστά μας και θα πρέπει να δώσουμε στα προβλήματα αυτά συνολικές απαντήσεις. Οι πολιτικές που αντιμετωπίζουν την περιπλοκότητα αυτή θα πρέπει να είναι συστημικές πολιτικές. Αν ο καθένας προσπαθήσει να δώσει μεμονωμένες απαντήσεις επί τη βάση των ιδίων αυτού συμφερόντων, τότε θα έχουμε όλοι να χάσουμε. Εγώ θέλω να υπάρχει μια ισχυρή γεωργία, μια ανταγωνιστική γεωργία και η εργασία των γεωργών να αναγνωρίζεται σαν σημαντική και χρήσιμη. Θέλω ένα περιβάλλον σωστό και προστατευμένο προς όφελος όλων. Θα κάνω ό,τι μπορώ από πλευράς μου προς την κατεύθυνση αυτή και νομίζω ότι και εσείς θα στηρίξετε την προσπάθειά μου. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Grazie. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Ευχαριστώ λοιπόν τον Γιάννη Σποτότσκι για αυτά που μας είπες. Είναι πολύ σημαντικά για μας και σε ευχαριστούμε. Ήταν σαφή αυτά τα οποία μας είπε, σαν Επίτροπος Γεωργίας και έδειξε την ευαισθησία που έχεις απέναντι στη Γεωργία και για την οποία σε ευχαριστούμε. Όλοι επιθυμούμε μια κοινή αγροτική πολιτική πιο πράσινη θα θέλαμε όμως αυτή η μεγαλύτερη θα έλεγα αναγνώριση να γίνει ε, στόχος χωρίς να περιπλακεί η ζωή των γεωργών μας. Θα πρέπει αυτό το πρασίνισμα σε εισαγωγικά να είναι μια πραγματική ευκαιρία και όχι μια χειροτέρευση της γραφειοκρατίας. Λοιπόν, ξεκινάμε τη συζήτηση. Έχουν ήδη γραφτεί πάρα πολλοί συνάδελφοι. Θα ξεκινήσω φυσικά δίνοντας το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Ντες, και μετά θα ακολουθήσουν όλοι όσοι έχουν ζητήσει το λόγο, αλλά προσπαθήστε να σεβαστείτε το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε που βρεθήκατε σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας και νομίζω ακούγοντας τις ε, θέσεις σας ότι αν βρούμε τους σωστούς, ε, τις σωστές οδούς και επιλέξουμε και τα σωστά μέσα δεν θα απέχουμε πολύ ε, οι θέσεις μας. Υπάρχει πάντο μία διαφορά μεταξύ πολιτικής για το περιβάλλον και πολιτικής γεωργίας, αλλά εγώ πάντα λέω ότι τους ίδιους στόχους θέλουμε να πετύχουμε, η ευρωπαϊκή γεωργία δηλαδή, να να καταστεί πιο βιώσιμη από ό,τι είναι. Εγώ ποτέ, κύριε Επίτροπε, δεν έχω δει πιο περιβολητικά φιλική γεωργία από αυτή που έχουμε σε κάποιες ε, περιοχές στην Ευρώπη. Σαφώς και υπάρχουν ελλείμματα και θα πρέπει να επέμπουμε για να καλυφθούν αυτά τα χάσματα. Και είπατε πολύ σωστά ότι η γεωργία δεν θα πρέπει να τιμωρηθεί. Θα πρέπει αντίθετα να ανταμείψουμε εκείνους που ήδη προστατεύουν το περιβάλλον. Και εδώ έχω ένα μεγάλο πρόβλημα στην έκθεσή μου. Μιλήσατε για τον πρώτο πυλώνα. Εγώ διαπιστώνω το εξή στην Ευρώπη επί του παρόντος. Κάνουμε πληρωμές ε, εξίσωση στον πρώτο πυλώνα βάσει ιστορικών πληρωμών μεταξύ 5 ευρώ ανά εκτάριο και πάνω από 600 ευρώ. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να πρασινίσει επί της αρχής ε, ο πρώτος πυλώνας όταν ε, ε, μία χώρα λαμβάνει 50 ευρώ ανά εκτάριο θα πάρει 15 και άμα είναι 600 τα ευρώ που παίρνει τώρα θα πρέπει να γίνουν πόσα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει δικαιοσύνη σε αυτήν την μεταρρύθμιση. Κάτι άλλο κύριε Επίτροπε πολύ σημαντικό κοίταξα τα στατιστικά στοιχεία για την ανάπτυξη των γεωργικών παραγωγών από το 76 μέχρι το 2008. 32 χρόνια στο χρονικό αυτό πλαίσιο στην Ευρώπη η παραγωγή δημητριακών ανέβηκε 1%. Όχι 1% ετησίως, 32 έτη σε άλλες αγροτικές περιοχές η αύξηση αυτή ήταν 200%, στην Ασία ήταν 100% η αντίστοιχη αύξηση και αν κινδούμε μια άλλη στατιστική, παραγωγή κρέατος στην Ευρώπη, 6% αύξηση, 307% η αύξηση αντίστοιχη στην Ασία. Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία, κύριε Επιτροπέ, θα πρέπει να τα έχετε υπόψη όταν εξετάζουμε ενδεχόμενα μέτρα για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη για να μην υπάρχει μεταγκατάσταση από την Ευρώπη σε άλλες αγροτικές περιοχές, γιατί αν συμβεί αυτό θα βλάψουμε και την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία του κλίματος και την προστασία των ζώων. Ξέρετε, κύριε Επίτροπε, ότι σε άλλες ε, γεωργικές περιοχές δεν υπάρχουν αντίστοιχα μέτρα και αντίστοιχες σκέψεις όπως στην Ευρώπη για την προστασία των ειδών αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε την ε, παραγωγή στην Ευρώπη γιατί δεν θέτουμε μόνο... Κοιτάξτε, δεν είναι ότι μόνο στην Ευρώπη έχουμε τις ανησυχίες που έχουμε, θα πρέπει να φροντίσουμε να βρούμε σωστή ρύθμιση. Και αν προέρχεστε από αγροτική περιοχή, θα ξέρετε ότι οι γεωργοί κερδίζουν καλύτερα όταν πείθονται ότι είναι σωστά τα μέτρα που τους επιβάλλονται. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να πετύχουμε, να συμμετάσχουν και οι ίδιοι οι γεωργοί. Κοιτώντας την Ευρώπη, γιατί ήμουν πρόσφατα στην Φιλανδία και πέταξα από το Ελσίνκι και είδα κάποια μέρη της Φιλανδίας και σκέφτηκα Μα τι να πρασινίσει παραπάνω στη Φιλανδία. Έχουν τόσα πολλά πράσινα στοιχεία που δεν μπορώ να επιβάλλω οτιδήποτε καινούργιο στην γεωργία, στους γεωργούς στη Φιλανδία και ξέρω άλλες περιοχές στην Ευρώπη όπου χρειάζεται να αναλυφθούν μέτρα. Ε, θα πρέπει να γίνει λοιπόν έντονη διαφοροποίηση, να κοιτάξετε τα αριθμητικά στοιχεία για τα 27 κράτη-μέλη, γιατί υπάρχουν κράτη-μέλη στην Ευρώπη όπου 40% και πάνω των ε, γεωργικών ε, εσόδων δαπανώνται για περιβαλλοντικά μέτρα. Και σε άλλες χώρες είναι 1% το ποσοστό αυτό. Έμα, πρώτα θα πρέπει να προσέξουμε και να φροντίσουμε να προστατευτεί το περιβάλλον όπου δεν προστατεύεται ακόμα επαρκώς. Γι' αυτό λοιπόν να κοιτάξουμε την προστασία του εδάφους, του ύδατος και σε ό,τι αφορά την προστασία του κλίματος θα πρέπει να φροντίσουμε μεταξύ των κρατών μελών να, υπάρχουν, να υπάρχει ισότητα και να μην υπάρχουν στρεμπλώσεις του ανταγωνισμού. Μιλήσατε με σαφήνεια κυρία Επίτροπε και μιλήσατε για, την για το διαρκές πρασίνισμα κοιτώντα τι γίνεται στη Γερμανία, στη χώρα μου. Στη Γερμανία Μέχρι το 2013 από τις πληρωμές εξισορρόπησης του πρώτου πυλώνα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανώνται για την μετατροπή ε, γεωργικών επιφανειών σε πράσινες επιφάνειες. Δηλαδή για τις πράσινες ε, επιφάνειες ε, δίδονται οι ίδιες πληρωμές όπως και για τις αγροτικές επιφάνειες ακριβώς οι ίδιες. Οι χώρες οι οποίες έχουν σημειώσει ήδη πολύ καλές επιδόσεις, δεν μπορούμε να απαιτήσουμε να επιβαρυνθούν με επιπρόσθετα μέτρα, τα οποία δεν έχουν ε, εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη. Ακόμα και αν συμφωνώ με αυτά, και θα χαρώ σε περίπτωση που έχουμε μία προσωπική κατηδίαν συζήτηση να μιλήσουμε και για την πολλαπλή συμμόρφωση. Γιατί πολλοί αγρότες δεν καταλαβαίνουν, για παράδειγμα, ότι οι έλεγχοι για την πολλαπλή συμμόρφωση έχουν επιπλέον κυρώσεις. Εδώ υπάρχει ένα σαφές ειδικό δίκαιο, μια ειδική νομοθεσία. Αν υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας αυτής, εντάξει να υπάρχουν κυρώσεις. Να μην υπάρχουν όμως διπλές κυρώσεις. Εγώ συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή, δυνατή γεωργία και να σκεφτείτε και το εξή, κύριε Επίτροπε. Η λέξη βιωσιμότητα προέρχεται από τον δασικό και γεωργικό τομέα. είναι αλλού δεν ε, υπήρχε αυτή η λέξη. Πάντα σε αυτές τις οικογένειες ο σκοπός ήταν να δίδονται στις, στις ε, επερχόμενες γενιές τα δάση και οι γεωργικές εκτάσεις στην ίδια κατάσταση που τα είχαν πάρει από του πατέρες τους. Ελπίζω λοιπόν να είναι καλή και η συνεργασία για να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται στον τομέα της γεωργίας. Ευχαριστώ Άλμπερτ. Ο κύριος Παπαστάμκος. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο για την ε, ενημέρωση που μας έκανε σήμερα και για την ε, προσέγγιση του φακέλου ε, μέλων της ΚΑΠ από μια άλλη σκοπιά. Ε, συμφωνώ απόλυτα μαζί του ότι χρειάζεται πράγματι η επανάσταση της κοινή λογικής, η επανάσταση του αυτονοήτου, ε, θα έλεγα. Αλλά σε ό,τι αφορά την, ε, τις προσδοκίες για την ανακατανομή των άμεσων ισχύσεων και ό,τι αυτό συνεπάγεται, θέλω να πω στον καλό συνάδελφο, στον κύριο Ντές, ότι είναι διαφορετικό να είναι κανείς γεωργό στην Ευρώπη ε, με 50 εκτάρια και να είναι γεωργό, κατ' επάγγελμα μάλιστα στην Ευρώπη με 2 εκτάρια. Επομένω υπάρχει και ένα άλλο κριτήριο κύριε Ντές. Πέρα από την έκταση των εκταρίων υπάρχουν και οι δικαιούχοι και τι πραγματικά ε, απολαμβάνουν ως άμεσες ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό απλώς ε, δεν είναι η ώρα να το αναλύσω αλλά πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Ε, κύριε Επίτροπε, ασφαλώς και η διατήρηση των θεμελίων της ζωής είναι μια οικουμενική εντολή. Έχει έναν οικουμενικό χαρακτήρα και δεν έχει χρώματα, αλλά ε, αναγνωρίζω πλήρως το στόχο για πρασίνισμα, τον φιλόδοξο στόχο της κοινή αγροτικής πολιτικής, όμως υπάρχει και μια άλλη διάσταση της κοινή αγροτικής πολιτικής, η εξωτερική δηλαδή η οικονομική γεωγραφία της κοινή αγροτικής πολιτικής, δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο, υπάρχει το παγκόσμιο ανταγωνιστικό πεδίο. Και αν εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρήσουμε, και ορθώς είναι θεμητός ο στόχος, σε περαιτέρω πρασίνισμα, αλλά άλλες ανταγωνίστρες δυνάμεις ε, υπολείπονται σημαντικά, τότε προσθέτουμε ένα ακόμη ανταγωνιστικό μειονέκτημα στην Ευρωπαϊκή ε, Γεωργία. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη επίσης δεν ακούω, φιλόδοξοι στόχοι απαιτούν και τα επαρκή ε, χρηματοδοτικά μέσα. Ε, δηλαδή μπορούμε να θέτουμε φιλόδοξους στόχους και αύριο μεθαύριο ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ελληματικός. Δηλαδή την ώρα που φορτώνουμε εντό εισαγωγικών την κοινή αγροτική πολιτική με μια νέα αποστολή, όπως είναι αυτή της οικολογίας, δεν μπορούμε να αφήνουμε τις δημοσιονομικές προοπτικές σε επίπεδο ανεπαρκές. Ε, αναφερθήκατε πολύ σωστά και τελειώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε στα μέτρα που έχει ήδη προτείνει η Κομισιόν, στην αμυψισπορά δηλαδή, την, ε, επαναλαμβάνω, αμυψισπορά, την οικολογική αγρανάπαυση, στους μόνιμους βοσκότοπους και στη φυτική κάλυψη. Αυτά, στη δική μου αξιολογική κλίμακα, απαντούν σε ένα τοπίο, σε μια κλιματική πρόκληση που αφορά την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη. Η κλιματική όμως ε, πραγματικότητα στον Ευρωπαϊκό Νότο είναι διαφορετική. Και πρέπει να ληφθεί και αυτή η υπόψη στις προτάσεις της, της Κομισιόν. Ε, και πράγματος χάρη δεν είναι... Γιατί να μην συμπεριλαμβάνεται η διατήρηση των αμπελώνων, των οπορώνων και των ελαιώνων σε καλή ε, βλαστική κατάσταση. και θα ήθελα τη θέση σας επ' αυτού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Grazie, grazie Επίτροπε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και που θέλετε να διεξάγουμε διάλογο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο τομέας, ο περιβαλλοντικό και η γεωργία να συνεργαστούν στενά. Και χαίρομαι λοιπόν που ξεκινήσατε αυτή την κοινή πρωτοβουλία γιατί επί τη ουσία, νομίζω ότι συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι πρέπει να ασκηθεί τέτοια γεωργική απολυτική που να μην έρχει σε αντίθεση με την περιβαλλοντική πολιτική. Και ότι και η γεωργία θα πρέπει να συμβάλλει στον προορισμό της αλλαγής του κλίματος. Και στο σημείο αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Δεν νομίζω ότι το ποσοστό της γεωργίας βρίσκεται στο 10% μόνο. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο υψηλό το ποσοστό αυτό. Για παράδειγμα, μέσω της εισαγωγής ε, ζωοτροφών που έχουν παραχθεί σε χώρες που δεν ε, ελέγχουμε εμείς. Και όλα αυτά θα πρέπει να λεφτούν υπόψη στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο, χωρίς να λαμβάνονται ακόμα υπόψη. Ε, θα ήθελα λοιπόν να πω ότι στην γεωργική πολιτική η αρχή του αμείβουμε αντί να τιμωρούμε είναι πολύ σημαντική. Δεν θέλουμε λοιπόν θέλουμε να ε, ενισχύσουμε στο τελική ανάλυση τους γεωργούς αυτούς που ε, προστατεύουν τον περιβάλλον και θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει διαφοροποίηση. Σε κάποιους τομείς υπάρχει μια τάση βιομηχανοποίησης και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό και θα πρέπει να δράσουμε. γιατί αυτή η περιβαλλοντική, αυτή η βιομηχανοποιημένη γεωργία προκαλεί πρόβλημα. Θεωρούμε λοιπόν ότι χρειάζεται βιώσιμη, διαρκή πίεση για να αλλάξει κάτω, κάτι στη γεωργική πολιτική, να δίνουμε κίνητρα ε, για να ανταμείβουμε τις γεωργικές πρακτικές που επιθυμούμε. Ένα άλλο θέμα που ήθελα να αναφέρω είναι το εξής. Το θέμα των βιοκαυσίμων. Νομίζω ότι στη στοχοθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την ε, βιομάζα υπάρχουν λανθασμένοι στόχοι. Και βρισκόμαστε λοιπόν σε μια αντίφαση μεταξύ, σε μια σύγκρουση μεταξύ της παραγωγής τροφίμων και την παραγωγή βιοκαυσίμων, η οποία δεν είναι αρκετά ε, βιώσιμη. Υπάρχουν λοιπόν ανάγκη βελτίωσης ε, της πολιτικής αυτής. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι θα πρέπει να προάγουμε την γεωργία σε περιοχές που βασίζονται σε λιβάδια. Θα πρέπει να είναι αυτό βασικό στοιχείο της ε, πολιτικής, της μεταρρύθμισης γεωργικής πολιτικής. Και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα ε, που διεξάγεται ο διάλογος αυτός για να διατυπώσουμε τους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής και της γεωργικής πολιτικής και να μην καταλήξουμε σε μια τεχνητή, αν θέλετε, σύγκρουση. Νομίζω ότι η καινούργια αγροτική πολιτική μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή μόνο αν υπάρχει υποστήριξη από πολλές ε, δημόσιες ομάδες για μια δίκαιη γεωργία και για τη δαπάνη των ε, κοινών κονδυλίων. Γιατί και αυτό θα παίξει πολύ βασικό ρόλο στη μερατική γεωργική πολιτική. Grazie Martin, Mark Tarabella. Ο Μάρκ Ταραμπέλα. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να αναφερθώ στις παλιές σας αγάπες, δηλαδή την πολιτική έρευνα, καθότι υπήρξατε αρμόδιος ε, μεταξύ του 2004-2009 αρμόδιος επιτρόπος για την ενέργεια. Και ο Φιλίπ Μπισκέ, ο προκάτοχό σα, αλλά και εσεί ο ίδιο, έχετε συνεισφέρει σημαντικά για, να, ε, για τι αντρέ γραμμέ του 7ου προγράμματο έρευνα και ανάπτυξη, που είχε μία από τι προτεραιότητέ του τη γεωργία. Τώρα λοιπόν βλέπουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους, οποίους ε, αναφέρατε, βιοπικιλότητα, διαχείριση εδαφών ε, και υδάτων, ε, η παγίδευση του άνθρακα που αναφέρατε, αλλά και η εξάρτηση από φυτικές πρωτεΐνες και καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Θα ήθελα να μου πείτε, η έρευνα μέσω του 7ου προγράμματος ε, πλαισίου. Ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει βέβαια πάντοτε ε, και εν ώψη του να σεβόμεθα και το περιβάλλον. Δηλαδή στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου πώς μπορούμε να εντάξουμε την έρευνα, να τη διαρθρώσουμε και στο πλαίσιο και της κοινή γεωργικής πολιτικής. José Κύριε Επίτροπε, Ήταν ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε, επικοδομητικά ήταν και λογικά. Αλλά ένα μικρό παράπονο έχω. Βλέπουμε τον επίτροπο μετά τον άλλο, τρεις επίτροποι νομίζω θα έπρεπε να είναι παρόντες και να μιλούν με μια φωνή γεωργία, περιβάλλον, κοινων... ε, καταναλωτές υγεία. Γιατί όλα αυτά είναι ένα σύνολο αυτά τα θέματα αλλά βλέπουμε μια σαλαμοποίηση παρόλα αυτά αυτών των τρών. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Είπατε ότι έχουμε πραγματικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Αυτό δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα. Βλέπουμε για τις μέλισσες ότι σχεδόν δεν έχουν μέλλον, αυτό είναι πραγματικότητα, αλλά θα πρέπει να δείξουμε και να κατονομάσουμε τους υπευθύνους, που είναι η πετροχημική βιομηχανία, είναι τα, παρα, τα παρασιτοκτόνα, είναι οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις αυτή τη συζήτηση, πρέπει να σταματήσει αυτό. Δεν θα έχουμε πράσινη κοινωνική πολιτική αν τα φυτοφάρμακα και οι γενετικώ τροποποιημένοι οργανισμοί συνεχίζονται να, ε, συνεχίζουν να έχουν τη στήριξη που έχουν. Αυτό πρέπει να είναι σαφέ. Τώρα, να σας πω κάτι άλλο σε σχέση με το θέμα τη αγορά. Δεν θα πρασινίσει η ΚΑΠ με ενισχύσει και μόνο με ενισχύσει. Οι αγρότες ζουν κυρίως από την αγορά. Άρα είναι προφανές ότι θα πρέπει να αμείβονται οι αγρότες για τη δουλειά τους. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση ώστε να μπορούν οι αγρότες να έχουν πρακτικές που θα τους επιτρέψουν να διατηρήσουν την απασχόλησή τους. Αν έχουμε αγώνα για όσο το δυνατόν πιο χαμηλές τιμές για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο γεωργοδιατροφικό τομέα, είναι προφανές ότι δεν θα έχουμε κάποιοι που θα σέβεται το περιβάλλον, Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πραγματική αντίφαση. Γι' αυτό και διαφωνώ με τη λογική του ανταγωνισμού. Έχουμε φτάσει πλέον στα άκρα. Αν ο κύριος Άλμπερτ Ντες μας λέει ότι δεν υπάρχει πια πρόοδος, πράγματι δεν υπάρχει γιατί έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο πια παραγωγικότητας που σήμερα ε, το κέρδος παραγωγικότητας για τον πλανήτη είναι στο χώρο, στους χώρες του Νότου κυρίως. Γιατί να αυξήσουμε, δεν έχει νόημα να αυξήσουμε την παραγωγή σε εμά, ενώ στο Νότο δεν έχουν τι να παραγάγουν και κάνουμε dumping στην παραγωγή. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια. Και τελευταίο σημείο για την αγορά, εάν πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε πιο πράσινη την ΚΑΠ, πολύ καλά, συμφωνώ. Αλλά η πολλαπλή συμμόρφωση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ε, αυστηροί σε ό,τι αφορά τα πρότυπα και τους κανόνες εισαγωγής. Έχουμε θέμα στον ΠΟΕ. Δεν θα πρέπει η Ευρώπη να συνεχίσει να θέλει να ε, χρησιμοποιεί τη γεωργία ως μια μεταβλητή προσαρμογή στην οποία ουσιαστικά παραχωρούμε στους άλλους τομείς. Πρέπει να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστώ ευχαριστω e Ευχαριστώ, Επίτροπε, και εγώ θα ήθελα να σα καλωσορίσω εδώ στην Επιτροπή μα, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών, η Γεωργία και το Περιβάλλον φαίνεται ότι αποτελούν ε, ασύμβατες έννοιες, τουλάχιστον αυτό ήταν στο παρελθόν, ίσως και αντιφατικές. Θυμάμαι ότι όταν ξεκίνησα την καριέρα μου ε, στο Υπουργείο μάλλον ε, Γεωργία στην Πορτογαλία, χρησιμοποιούσαμε τον δείκτη ένταση χρήσης ε, σε ό,τι αφορά τους γεωργούς για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνταν για να βελτιώσουν τη γεωργική παραγωγή. Νομίζω ότι τα τελευταία 20 χρόνια είδαμε ότι το γεωργικό περιβάλλον, μάλλον η γεωργία και το περιβάλλον κατέστησαν έννοιες συμπληρωματικές, όχι πλέον αντιφατικές. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθήσουμε και στο μέλλον. Οι συζητήσεις οι οποίες διεξάγονται στην παρούσα φάση για το ε, μέλλον της ΚΑΠ, αυτό έχουν ως σκοπό για την προστασία και το σεβασμό του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να προστατεύεται και το εισόδημα των γεωργών και να διασφαλίζεται ότι η γεωργία θα αποτελεί μια βιώσιμη απασχόληση και στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκ παραλίλου. Ασφαλώς και θέλουμε να προστατεύσουμε το έδαφος, τη βιοπικιλότητα, την ποιότητα του ύδατος, ε, τα δάση. Το ενεργειακό ισοζύγιο θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε ό,τι αφορά την προστασία μάλλον την ε, μείωση της αλλαγής του κλίματος, όλα αυτά θα πρέπει να λεφθούν υπόψη στην ΚΑΠ. Και όλο και πιο πολύ βλέπουμε ότι η πιο πράσινη ΚΑΠ με την κατάλληλη χρηματοδότηση αποτελεί μια επιταγή πραγματικά για το μέλλον των πολιτών μας. Δεν επιχειρούμε απλά να ικανοποιήσουμε τους πολίτες και τις ενστάσεις τους. Όχι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τους γεωργούς και τους πολίτες μας στο μέλλον. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο κόσμος μας θα είναι προστατευμένο στο μέλλον. Η ομάδα των σοσιαλιστών εξετάζει την ΚΑΠ και όλες τις περιβαλλοντικές και αγιεργικές πτυχές και είμαστε πραγματικά δεσμευμένοι για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε μια συνοχή, μια συνέπεια και μια αναλογικότητα στις αντιδράσεις μας. Σε ό,τι αφορά την έκταση του προβλήματος, θα πρέπει να καταδείξουμε, ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει σωστή αποζημίωση επίσης των Γεωργών. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που βρίσκεστε εδώ μαζί μας και μας παρουσιάζετε αυτό το σημαντικό θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε στο μέλλον και από άλλη οπτική γωνία. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και που με εντυπωσιάζει γενικότερα στην όλη συζήτηση για το πρασένισμα της γεωργίας είναι το γεγονός ότι κι εσείς σήμερα δεν μιλήσατε για το μέσο, το μέσο κατεξοχήν ε, για το πρασίνισμα της ε, γεωργίας, για τα εθελοντικά μέσα που υπάρχουν στο δεύτερο πυλώνα της γεωργικής πολιτικής, υπάρχουν εδώ και 20 χρόνια, υπάρχουν μια σειρά παραδειγμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία καταδεικνύουν ότι το μέσο αυτό λειτουργεί πραγματικά θαυμάσια. Και υπάρχουν, όπως είπε και ο εισηγητής Άλμπερτ Ντάς, υπάρχουν άλλες περιοχές όπου τα μέσα αυτά δεν λειτουργούν καθόλου γιατί δεν προσφέρονται από τις χώρες σχετικά προγράμματα ή δεν τα αποδέχονται οι γεωργοί. Και η σχέση μεταξύ των κρατών που κάνουν τα πιο πολλά και των κρατών που κάνουν τα πιο λίγα είναι 1 προς 20 περίπου. Η αναλογία. Και νομίζω ότι όταν μιλάμε για μια πιο πράσινη γεωργία θα πρέπει να μιλάμε για, τα, για τις χώρες όπου έχει νόημα. Ένα παράδειγμα από την περιοχή μας, για παράδειγμα, στις Άλπεις. Όταν εξηγεί κανείς τις σκέψεις του και τα όσα είπατε πριν από λίγο για την απαγόρευση, μάλλον για την ε, το υποχρεωτικό πρασίνισμα με της μεταφοράς στην πρώτο πυλώνα. Αυτό τι σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε πλέον να χρηματοδοτούμε τα μέτρα αυτά ως ε, μέτρα εθελοντικά στην δεύτερο πυλώνα και θα συμβεί αυτό που είπε ο εισηγητής, ότι υπάρχουν κάποιες ε, περιοχές όπου έχουν γίνει κάποιοι ιστορικοί υπολογισμοί Άρα οι γεωργοί θα χάσουν το αγροτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα και δεν θα λάβουν τίποτα και άρα θα τα καταλήψουν. Όχι μόνο λοιπόν δεν θα έχουμε πετύχει τίποτα, αλλά θα έχουμε και να, κάνει και ένα βήμα προς τα πίσω. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ όταν μιλάμε για το πρασένισμα θα πρέπει να κοιτάξουμε τι συμβαίνει ήδη σήμερα στα κρατημέλη και ποια είναι η κατάσταση, το σημείο κίνησης. Θα άξιζε τον κόπο να σκεφτούμε μήπως η σαφής αύξηση των προγραμμάτων τα περιβάλλων θα είχε ίσως πιο πολλά αποτελέσματα από ότι κάτι εθελοντικό. Γιατί υπάρχουν παραδείγματα στην Ευρώπη τα οποία θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε βέλτιστα παραδείγματα και από τα οποία θα μπορούσαμε να διδαχτούμε. Ευχαριστώ. Grazie Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι. Θα ήθελα να εκφράσω την βαρέσκειά μου γιατί ξαφνικά αρχίσαμε να μιλάμε για τη γεωργία σαν φυσικό πόρο και να εντάσσουμε υποχρεωτικά πλέον την γεωργία στο θέμα του περιβάλλοντος. Εμείς πάντα υποστηρίζαμε ότι η γεωργία και η εκμετάλλευση των βασών ήταν κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για την κοινωνία μας συνολικά. Κάποιοι βέβαια υποστήριζαν ότι η γεωργία ήταν βασικά βάρος για την κοινωνία. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτή η λανθασμένη αντίληψη οφειλόταν σε λανθασμένα ευρωπαϊκά μέτρα. πρέπει νομίζω κύριε Επίτροπε να ξεκινήσουμε πλέον να βλέπουμε με διαφορετικό τρόπο το θέμα της γεωργίας και του περιβάλλοντος. Με ενιαίο τρόπο η γεωργία εντάσσεται στο περιβάλλον και ο καθένας μας έχει ένα θέμα το οποίο τον ενδιαφέρει μεμονωμένο και θα πρέπει να τα συνδυάσουμε αυτά για να καταλήξουν σε συνολικές προτάσεις. Ένα από τα θέματα τα οποία βρίσκω πάρα πολύ σημαντικά είναι η σύνδεση ανάμεσα στις περιοχές της υπαίθρου και στις περιοχές με υψηλές αστικές συγκεντρώσεις. Ξέρουμε ότι υπάρχει ουσιαστικά μια αύξηση του πληθυσμού στον κόσμο γενικότερα. Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχει και μια τάση ε, πληθυσμιακών ροών προς τις πόλεις, τις αστικές περιοχές. Είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε όμως ε, περιοχές κατοικίας και στην Ήπεθρο, περιοχές τις οποίες να υπάρχουν σύγχρονα μέσα ε, επιβίωσης, διαβίωσης, συγγνώμη, έτσι ώστε να αποτραπεί η φυγή προς τις πόλεις και η απερίμωση ουσιαστικά των γεωργικών περιοχών η γεωργία την οποία έχουμε μπροστά μας λειτουργεί μόνο με λογικές παραγωγικές. Νομίζω ότι καθημερινά παράγουμε προϊόντα, τρόφιμα τα οποία μετακινούνται από την επαρχία στις πόλεις και η κατάσταση που δημιουργείται δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Είναι επιβαρυντική για το περιβάλλον. Δυστυχώς δεν υπάρχουν απαντήσεις ε, προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με τα θέματα των αποβλήτων, έτσι ώστε αυτά τα οποία μεταφέρονται στις πόλεις θα πρέπει ότι περισσεύει μετά από τη χρήση τους να επιστρέφουν στην περιφέρεια έτσι ώστε να υπάρχει μια αμφίδρομη θα έλεγα μορφή μεταφοράς ανάμεσα στις πόλεις και στην Ήπεθρο και να έχουμε την δυνατότητα χρήσης φυσικών λίπασμάτων και να διατηρήσουμε τα εδάφη σε καλή κατάσταση και τους υδάτινους πόρους και τη θάλασσα επίσης σε καλή κατάσταση. Διαρωτώ λοιπόν, μια τέτοια συζήτηση δεν σας ενδιαφέρει. Μια τέτοια συζήτηση δεν είναι απαραίτητη πριν πάρουμε τμηματικές αποφάσεις. Λαβία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να στραφώ προς τον Επίτροπο Ποτότσνικ, όχι τόσο σαν Επίτροπο υπεύθυνο για το περιβάλλον, αλλά σαν τμήμα του συνόλου των Επιτρόπων. Θα ήθελα να συζητήσω μαζί του ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το σύνολο της Επιτροπής γύρω από τον προϋπολογισμό που προορίζεται για την ΚΑΠ. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο. Στα πλαίσια των νέων δημοσιονομικών προοπτικών, ήδη εδώ και αρκετό καιρό, σχετικά με τις... Ε, έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στοιχεία και κάποια έγγραφα και μάλιστα είχε συζητηθεί και ένα non-paper το οποίο προέβλεπε σαφέστατη μείωση πιστώσεων προς την ΚΑΠ. Τώρα έχουμε και μία επιστολή η οποία μας έχει σταλεί από πέντε πρωθυπουργούς που ζητούν στα πλαίσια του Συμβουλίου να αποστηρώσουν τον νέο προϋπολογισμό και να το περιορίσουν σε αυξήσεις το πολύ 1%. Θα ήθελα λοιπόν να υπενθυμίσω σε όλους και στον Επίτροπο ότι η ΚΑΠ προβλέπεται από τις ιδρυτικές συνθήκες της Ένωσης είναι μία από τις βασικές πολιτικές της Ένωσης και είναι σαφές ότι δεν θα μπορούσαμε να διανοηθούμε ένα μέλλον της Ένωσης εάν δεν συνεχιστεί μία ισχυρή ΚΑΠ. Σήμερα εμείς ζητάμε από την ΚΑΠ ακόμα πιο σημαντικές παρεμβάσεις. Σήμερα από την ΚΑΠ ζητάμε εκτός από την εγγύηση της προμήθειας σε τρόφιμα, εκτός από την εγγύηση της ασφάλειας των τροφίμων, ζητάμε από την ΚΑΠ να σεβαστεί το περιβάλλον, να προστατεύσει το περιβάλλον, να παράγει αγαθά καθολικής ωφέλειας, ζητάμε συνεχώς όλα και περισσότερα. Και δεν μπορούμε λοιπόν από τη μία να τα ζητάμε όλα αυτά, να ζητάμε δηλαδή περισσότερα από τους γεωργούς και από την άλλη να τους υποβάλουμε όλο και πιο άδικα στην, στον διεθνή ανταγωνισμό γιατί έχουμε τα προβλήματα που έχουμε με τις υποανάπτυξη χώρες που μπορούν να εξάγουν και γεωργικά προϊόντα στην Ευρώπη και δεν μπορούμε ταυτόχρονα να μειώνουμε τους πόρους του αγροτικού τομέα. Γι' αυτό λοιπόν στα πλαίσια των νέων δημοσιονομικών προοπτικών και στα πλαίσια του νέου πολιετούς προγράμματος θα πρέπει να υπάρξει μια σαφέστατη κάλυψη των αναγκών από τις πιστώσεις. Εμείς έχουμε ήδη ψηφίσει ότι το νέο αυτό δημοσιονομικό πλαίσιο δεν μπορεί να προβλέπει λιγότερους πόρους για την κοινή αγροτική πολιτική. Ένα δεύτερο θέμα, δευτερεύον και κλείνω για δεν έχουμε χρόνο αναφερόμενη στη σχέση περιβάλλοντος και γεωργών. Τα είπε ο κύριος Ντες είπε ότι η κατάσταση στην Ευρώπη διαφοροποιείται πάρα πολύ. Υπάρχουν χώρες που δεν λαμβάνουν περιβαλλοντικά μέτρα, υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες όμως εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά και αφορούν τα μέτρα αυτά το 40% της γεωργικής παραγωγής τους. Φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Στην αρχική συζήτηση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαμε μιλήσει για το πρασίνισμα σε εισαγωγικά του πρώτου πυλώνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην, στο να γίνει το σύστημα πιο περίπλοκο. Και εσείς σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλετε να γίνουν πιο απλά τα πράγματα. Γιατί να μην περάσουμε σε μια μεγαλύτερη ομογενοποίηση του δεύτερου πυλώνα, έτσι ώστε ένα ποσοστό, μία ποσόστοση μάλλον του 20-30% των πιστώσεων που προορίζονται στον δεύτερο πυλώνα υποχρεωτικά να χρησιμοποιούνται για αγροοικολογικά μέτρα, απαλλάσσοντας τον πρώτο πυλώνα από περαιτέρω δεσμεύσεις και διευρύνοντας τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν τα νέα αυτά μέτρα. Ευχαριστώ Τζοβάνι Λαβία. Ναι, σας ευχαριστώ και χαίρομαι που ήρθατε και εσείς εδώ στην Ευρωπαϊκή μας σήμερα. Καταρχάς διαπιστώνω ότι είναι σωστό για τη γεωργική πολιτική και για την ε, περιβαλλοντική πολιτική οι αποφάσεις μας να λαμβάνονται υπόψη βάση ε, συγκεκριμένων περιστατικών και όχι βάση ε, θερμών εντάσεων και συναισθημάτων. Όχι, θα πρέπει να έχουμε σαφή και ακριβή στοιχεία προκειμένου να βασίσουμε σε αυτά την νομοθεσία μας. Κοιτώντας λοιπόν και βλέπουμε ότι θέλουμε μεγαλύτερη παραγωγή τροφίμων, αλλά θέλουμε και μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Να μην προκύψει μια αντίφαση μεταξύ των δύο αυτών παραγόντων. Και νομίζω ότι αν ε, θέλουμε πιο πολύ σύγχρονη τεχνολογία και πιο πολύ επιστήμη στον τομέα αυτό και πιο πολύ κατάρτιση στο γεωργικό τομέα, υπάρχει ε, δυνατότητα να αναπτυχθούν μέσα για να πετύχουμε αυτά που ε, επιθυμούμε. Προκειμένου να είναι συμπληρωματική αυτή η εξέλιξη και όχι αντιφατική. Και αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι να σταματήσουμε να λέμε ότι ε, είναι θέμα μεγέθους η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Δεν έχει να κάνει με το μέγεθος μιας επιχείρησης η προστασία του περιβάλλοντος. Το θέμα είναι τι κάνει ο Γεωργός με τα μέσα που έχει στη διάθεσή του. Αυτό, έχει, ε, αυτό είναι το πιο καθοριστικό στοιχείο. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε οι αποφάσεις μας να βασίζονται σε στοιχεία ακριβίας και όχι σε προκαταλήψεις. Αυτό να αποτελέσει τη βάση της μελλοντική γεωργίας. Και η γεωργία να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητη πλέον σε τέτοια ζητήματα. Abbiamo Daciana Sarbo e poi l'ultimo intervento Sarbo. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ένα είναι το θέμα που θέλω να θέσω. Η παραγωγή των βιοκαυσίμων είναι εδώ τίθεται και το θέμα βέβαια της αύξησης ε, της εκπομπής ε, διοξιδίου του άνθρακα. Ο στόχος αυτός του 10% για την χρήση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας στις μεταφορές, ιδιαίτερα τα βιοκαύσιμα μέχρι το 2020, θα μπορούσε να λειτουργήσει αρνητικά και να οδηγήσει σε αύξηση της εκπομπής καυσαερίων και όχι σε μείωση. Ευχαριστώ κυρία Σάρμπου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στο τέλος μια σύντομη ερώτηση προς τον Επίτροπο. Καρότο ή μαστίγιο. Όλοι προσπαθούμε να είμαστε όλοι κερδισμένοι, η γεωργία, κλιματική αλλαγή, βιοπικιλότητα κτλ. κτλ αλλά για να κινηθούν τα πράγματα, για να ε, κινηθεί αν θέλετε το γαϊδούρι ή θα το τιμωρήσεις ε, ή, ε, και θα του αφαιρήσεις πληρωμές στην περίπτωση της, των γεωργών ή μια θετική αντιμετώπιση, θετικά ερεθίσματα. Τι λοιπόν θεωρείτε, ποια είναι η απάντησή σας για το καρότο ή μαστίγιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ που πήρατε την πρωτοβουλία και καλέσατε τον αρμόδιο για το περιβάλλον επίτροπο, γιατί ε, ίσως είναι καλό σήμερα να κάνουμε αυτόν τον διάλογο για να βγούμε από αυτόν τον αγώνα, γιατί περί αγώνα πρόκειται μεταξύ γεωργίας, ε, περιβάλλοντος κτλ. Ε, πρέπει όλοι να συνεργαστούμε. Εσείς ε, δείξατε κύριε Επιτρόπε, ότι γνωρίζετε καλά τα, τα πράγματα στη Γεωργία, το αποδεικνύει και η διάδρομη σας μέχρι τώρα. Το θέμα είναι ότι έχουμε κάποια διοικητικά εμπόδια που είναι αποσυνδεδεμένα από τη γεωπονική πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Είπατε ότι και εσείς ότι θα θέλατε να έχουμε μια θετική στήριξη προς τη γεωργία σε θέματα περιβάλλοντος θα μπορούσατε να επεκταθείτε λίγο, να μας δώσετε κάποια παραδείγματα. Τι σκέψεις κάνετε σχετικά, πώς θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτή την πολιτική στήριξη και όχι πολιτική περιορισμών, αλλά να έχουμε και το ίδιο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ όλους. Νομίζω ότι ο Επίτροπος Γιάννης Ποτότσκι μας έδωσε ένα αισθαντανέ της κατάστασης και κάλυψε όλες τις ευαισθησίες των μελών της επιτροφής τους οποίους ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις τους. Έχετε το λόγο για να κλείσει η συζήτηση, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την συνεισφορά σας, τις ιδέες σας και που μου δίνετε την δυνατότητα να μιλήσω ελεύθερα να προσπαθήσω να εξηγήσω λίγο καλύτερα την κατάσταση της περιβαλλοντικής πολιτικής. Πώς τη βλέπω εγώ, κάτι το οποίο αποτελεί ουσιαστικά απλούστευση των πραγμάτων, πώς έβλεπα το θέμα πριν γίνω επίτροπος και πώς το βλέπω τώρα. Υπάρχουν πάρα πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το περιβάλλον. Λοιπόν, υπάρχει βάρος νομοθετικό δηλαδή, δεν υπάρχει θέμα. Έχουμε λοιπόν ένα σαφές νομικό σώμα εδώ, το οποίο κατά καιρούς αναθεωρούμε, αλλά η βασική νομοθετική ρύθμιση είναι σε ισχύ εδώ και καιρό. Χωρίς να θέλω τώρα να ξεκινήσω συζήτηση για την οδηγία, για την ποιότητα του εδάφους κτλ. Πάντως αυτή είναι η κατάσταση. Το θέμα είναι πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Κάθε βιομηχανική δραστηριότητα αναπτυσσόταν μόνη της και κανένας δεν ελάμβανε υπόψη το τι έκανε ο άλλος. Τελικά καταλήξαμε σε μία κατάσταση και βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, παραβιάσεις σε διάφορους τομείς, στον τομέα της προστασίας ε, του εδάφου, στον τομέα της προστασίας των υδάτινων πόρων και γι' αυτό αρχίσαμε να παίρνουμε νομοθετικά μέτρα λόγω ακριβώς των ανησυχιών που είχαμε ε, στον τομέα της υγείας και στον τομέα του περιβάλλοντος. Είχαμε προχωρήσει πάρα πολύ λοιπόν και αν θέλαμε να ελέγξουμε τα πράγματα έπρεπε να υιοθετήσουμε νομοθετικά μέτρα τα οποία από τη φύση τους ήταν αντιθετικά γιατί στην ουσία ζητούσε πάρα πολλές διορθώσεις στις υπάρχουσες δραστηριότητες και μάλιστα πολλές φορές επαναφορές προς τα πίσω. Το θέμα είναι τώρα πια να προβλέπουμε τα πράγματα αυτά πριν γίνουν. Αυτό έχει σημασία, να κατανοήσουμε ότι αυτό θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε σημαντικά προβλήματα στο μέλλον, μείζωνα προβλήματα, κάτι το οποίο είναι έτσι και αλλιώ προβλεπόμενο από την νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σχετική με την ΚΑΠ. Έχουμε την οδηγία πλαίσιο για τους υδάτινους πόρους. Είναι νόμος στην Ευρώπη. Πρέπει να εφαρμοστεί από το 12. Μία από τις απαιτήσεις της οδηγίας αυτού πλαισίου είναι ότι όλες οι χώρες από το 2015 θα πρέπει να έχουν τους υδάτινους πόρους τους σε εξαιρετική κατάσταση. Αν το λάβουμε αυτό από τώρα υπόψη, όταν ασχοληθούμε με άλλα θέματα στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και της γεωργίας ακόμα περισσότερο, αν δεν αναφερθούμε εμείς να συμφωνούμε τα μέτρα που θα πάρουν με τις ρυθμίσεις που είναι σε ισχύ, θα κάνουμε πολύ σημαντικά λάθη. Δεν θα σεβαστούμε τις πολλαπλές συμμορφώσεις. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι σε 4-5 χρόνια θα έχουμε προβεί σε παραβιάσεις οι οποίες θα είναι εναντίον των επιτρεπομένων πρακτικών και θα προκαλέσουν αντίμετρα οδυνηρά και δεν είναι σωστός αυτός ο τρόπος προόδου. Πρέπει να αποτρέψουμε λοιπόν κάποιες από τις συγκρούσεις που βλέπω να δημιουργούνται στο μέλλον. Αυτές λοιπόν οι ολοκληρωμένες πολιτικές είναι αυτές που είπα. Εγώ δεν θα ήθελα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και το περιβάλλον σήμερα. Ε, είπαμε ότι Μιλάμε για 2,3 δις σε μία επταετή περίοδο. Δεν μιλάμε και για κανένα πολύ σημαντικό προϋπολογισμό. Εγώ δεν ζητώ να αυξήσω το προϋπολογισμό αυτό. Το θέμα είναι να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία μπορούμε. Να διασυνδέσουμε τις πολιτικές μας, να βάλουμε τις πολιτικές μας στην πολιτική γεωργίας και αντίστροφα και έτσι θα πετύχουμε δύο στόχους ε, με μία προσπάθεια. Τώρα τα κράτη-μέλη, αναφερθήκατε πολύ στα κράτη-μέλη τα οποία κάνουν τα πράγματα που πρέπει να κάνουν πολύ καλύτερα από άλλα κράτη-μέλη. Προφανώς, αυτό είναι γεγονός. <clears throat> Και υπάρχουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες πρέπει να προκαλέσουν την προσοχή μας. Οι χώρες οι οποίες σήμερα, μέχρι σήμερα, είναι θα έλεγα οι καλύτεροι μαθητές στην χρήση του δεύτερου ιδιαίτερα πυλώνα ε, σκέφτονται να επεκταθούν οι ρυθμίσεις αυτές και στον πρώτο πυλώνα. Εδώ η λογική μου είναι απλή. Καταρχάς είναι υποχρεωτικό για κάθε γεωργό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι εγώ αν συλλέγω, ένα, αν παίρνω ένα ευρώ από τον καθένα από σας στο τέλος, θα έχω στην Ευρώπη 500 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι σημαντικό. Αν πάρουμε λοιπόν λίγα χρήματα από όλους τους γεωργούς οι οποίοι θα πρέπει να υπακούσουν ως προς αυτό, τότε θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε τα πράγματα. Και αυτό δεν είναι εναντίον της λογικής λειτουργίας του δεύτερου πυλώνα. Εγώ διευκρίνησα γιατί ο δεύτερος πυλώνας πρέπει να λειτουργήσει με καλύτερο τρόπο στο μέλλον. Αλλά νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να κάνουμε κάποια πρώτα μικρά βήματα γιατί τώρα έχουμε την ευκαιρία. Ποτέ δεν ήμασταν τόσο κοντά σε κάτι το τόσο σημαντικό. Αν δει κανείς τα θέματα αυτά, καθένας βέβαια τα βλέπει με διαφορετικό τρόπο, αλλά τα θέματα των υδάτινων πόρων και της βιοπικιλότητας. Η βιοπικιλότητα, μεγάλη υπόθεση για την Ευρώπη. Έχουμε την έκθεση του 2010 που λέει ότι χάνουμε με μεγάλη ταχύτητα και γι' αυτό οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πέρυσι υιοθέτησαν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για το μέλλον η στρατηγική της βιοπικιλότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δημοσιευθεί την 4η Μαΐου και θα καλύψει, καλύψει όλα αυτά τα θέματα εφόσον θέλουμε εμείς να αντιστρέψουμε αυτή την προϊούσα απώλεια της βιοπικιλότητας. Το ίδιο και για τους υδάτινους πόρους. Γνωρίζουμε όλοι ότι ένα από τα βασικά προβλήματα στο μέλλον είναι τα νερά. Εγώ είχα πάει την Παρασκευή στην Ελλάδα το 80%, πάνω από 80% του νερού των υδάτινων πόρων χρησιμοποιείται στη γεωργία. Είναι γεγονός αυτό. Δεν το κρίνω θετικό ή αρνητικό. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Οπότε δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ένα άλλο θέμα το οποίο έθεσε ο κύριος Ντέις πάρα πολύ σωστά. Πρέπει οι γεωργοί να κατανοήσουν και να συμμετέχουν στις προσπάθειες. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν θέλω να απομονώσω τους γεωργούς από την άλλη πλευρά και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας μόνοι μας από τη δική μας. Όχι, αυτό δεν θα δουλέψει ποτέ. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι πρώτον εκτιμούμε το τι είναι οι γεωργοί και τι δουλειά κάνουν οι γεωργοί. Μας παρέχουν τρόφιμα και παίζουν τον ρόλο τους αυτό πάρα πολύ καλά, όχι μόνο στον τομέα του περιβάλλοντος αλλά γενικότερα. Από την άλλη όμως, εφόσον συμφωνούμε ότι αν του 50% των γεών ελέγχονται από τους γεωργούς και αν συμφωνούμε ότι κάποιος θα πρέπει για λόγους βιοπικιλότητας να διαχειριστεί τα εδάφια αυτά, καλύτερα δεν θα ήταν να τα κάνουν αυτά οι γεωργοί παρά κάποιοι άλλοι, δηλαδή να κάνουν τη διαχείριση οι γεωργοί παρά κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, είναι απαραίτητο να γίνει αυτό και θα πρέπει να πληρωθούν από εμά για να μας παρέχουν αυτή την υπηρεσία κοινή ωφέλεια, η οποία δεν θα μπορούσε ουσιαστικά να γίνει αν δεν ήταν η Γεωργία εκεί που είναι σήμερα. Υπήρξαν επίσης και για τον προϋπολογισμό πολλές ερωτήσεις και τα μέτρα λιτότητας Νομίζω ότι δυστυχώς η κατάσταση στα δημοσιονομικά είναι αυτή που ξέρετε και η συζήτηση είναι πολύ δύσκολη. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Νομίζω ότι αυτή η πολλαπλή στρατηγική, η στρατηγική πολλαπλών επιπέδων για πολλαπλούς στόχους, στο τέλος είναι το μόνο πράγμα το οποίο θα έχουμε στη διάθεσή μας αν θέλουμε να καλύψουμε όσο περισσότερα προβλήματα έχουμε μπροστά μας. Θα είμαστε επίσης υποχρεωμένοι να δούμε και το θέμα των καινοτόμων τρόπων χρηματοδότησης. Αναπόφευκτο αυτό. Όταν ήμουν υπεύθυνο για τα θέματα της έρευνας, όπως είπε κάποιος από σας, ακόμα και εκείνη την εποχή, είχα υπογραμμίσει σαφώς ότι δεν είναι σωστό δεν είναι δίκαιο να συγκρίνει κανείς τις δαπάνες για τη γεωργία από τη μία και τις δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη από την άλλη. 5% για την έρευνα και την ανάπτυξη, ενώ για τη γεωργία μιλάμε για ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Λοιπόν, νομίζω ότι αν δεν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές θα πρέπει το ποσοστό για τη γεωργία να είναι πάντα υψηλότητα γιατί το σύστημα λειτουργίας και χρηματοδότησης το απαιτεί. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι θα πρέπει να κατανοήσουμε και εσείς φυσικά στην Επιτροπή Γεωργίας. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι όμως ότι πρέπει να προστατεύσουμε και τα άλλα συμφέροντα άλλων τομέων. Τώρα για το, η λογική του καρότου και του μαστιγίου. Η μέθοδος αυτή, η πολιτική αυτή, ακολουθεί αυτά τα οποία είπα στην, πρώτη, στην αρχή της παρουσίασής μου. Αν ακολουθήσουμε τη λογική της ολοκλήρωσης, περνάμε μέσα από τη λογική του καρότου. Αν μιλήσουμε για την απλή εφαρμογή των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τότε εκεί μιλάμε για το μαστίγιο. Υπάρχουν αρκετές χώρες σήμερα οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας. Θιούχα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Η αλλαγή αυτής της λογικής από το καρότο στο μαστίγιο είναι μια αλλαγή η οποία νομίζω θα αφελήσει τους Γιώργους συνολικά για την έρευνα και τι ρόλο μπορεί να παίξει η έρευνα. Όταν ήμουν υπεύθυνο για το πρόγραμμα Απλαίσιο, προσπαθήσαμε εμείς να διαμορφώσουμε την ερευνητική πολιτική μας έτσι ώστε να καλύπτει πολλαπλούς τομείς. Υπήρχε ένα σημαντικό τομέα, ένας από τους δέκα πυλώνες ήταν το περιβάλλον, αλλά τα βασικά γινόντουσαν βέβαια στην ενέργεια, στις μεταφορές, στις πρωτεσίλες κτλ. Ήμασταν πολύ πίσω, εν πάση περιπτώσει, από αυτό το οποίο θέλαμε να πετύχουμε, δηλαδή τη βιοοικονομία τη βασισμένη σε νέα γνώση. Είναι απαραίτητο λοιπόν να ληφθούν τέτοια μέτρα στο μέλλον. As you said, Bove, uh, sorry. Για σας κύριε Μπού. Here more commissioners. I think uh, εγώ δεν είμαι κατά της ιδέας για να υπάρξουν περισσότεροι επίτροποι δηλαδή. Αλλά αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω είναι να συνεργαστώ σε διμερές επίπεδο με όλους τους επιτρόπους με τους οποίους συνεργάζομαι και με τον επίτροπο Τσίολος έχουμε μία μόνιμη θα έλεγα συνεργασία και ακριβώς και η κοινή επιστολή που στείλαμε δείχνουν ότι δεν υπάρχουν διαφορές στην Επιτροπή. Δεν λέω ότι συμφωνούμε για τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά κάνουμε προσπάθειες και καταλήγουμε σε συμφωνίες. Δυνεπώς οι διαφορές υπάρχουν εκτός Επιτροπής, κυρίως στο Συμβούλιο και όχι τόσο στην Επιτροπή. Οι εμπορικές συμφωνίες και ο ΠΟΕ, προφανώς ο βασικό συστατικό της πολιτικής μας. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι σαν παράδειγμα στα πλαίσια της συμφωνίας με τη Μερκοσούρα. Εγώ πάντα ζήτησα να υπάρξουν σημαντικές ε, ε, ρήτρε προστασίας ε, των ρητρών, τις οποίες έχουμε συνάψει με τους συμβαλωμένους και συνεργαζόμαστε με τον Επίτροπο Τσίολος και τον Επίτροπο Ντεχούχτ για να κάνουμε επίσης και μελέτες βιωσιμότητας στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων. Όλα αυτά όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν μπορώ να σας δώσω κάτι περισσότερο. Είναι όμως θέμα το οποίο λαμβάνουμε υπόψη μας οι διεθνείς υποχρεώσεις μας. Για την προστασία... Anymore. Mr. Santos was that uh, uh, mentioned that, so I fully agree with that. I think it is a part which has. Δεν λέω σωστά το όνομά σα, κύριε Σάντου Καπούλα ε, για την προστασία του εισοδήματο των γεωργών. Είπαμε τα μέτρα που λαμβάνουμε. Τα εθελοντικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντο. εφόσον υπάρξει τελικά νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την περιοπτικότητα σε θείο και τα λοιπά των υδάτινων πόρων. Το θέμα δεν είναι αν θα ληφθούν θελοντικά μέτρα ή υποχρεωτικά μέτρα δεσμευτικά. Το θέμα είναι αν μπορούμε εκ των προτέρων να αντισταθμίσουμε με πληρωμές αυτούς οι οποίοι δεν θα εμπλακούν σε κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν από άμεσες παμοθετικές ρυθμίσεις για τις οποίες δεσμευόμαστε από τη συνθήκη να θέσουμε σε λειτουργία, σε εφαρμογή. Συνεπώς λοιπόν εγώ σε καμία περίπτωση δεν έχω εκφραστεί σε επίπεδο αρχής κατά των εθελοντικών ρυθμίσεων, αλλά όμως νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα εδώ Οι εθελοντικές ρυθμίσεις μας έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση η οποία δείχνει ότι διάφορα κράτη-μέλη δεν κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Για την κυρία Πόλσον, πράγματι κάνατε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια για την διατήρηση της ζωής και στις περιοχές της υπαίθρου. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αναφερθήκατε επίσης κύριε Πόλσον σε κάτι το οποίο είναι πολύ κοντά στις βασικές μου δραστηριότητες για τα θέματα των αποβλήτων που μπορούμε να έχουμε στην Ευρώπη. 179 κιλά αναπολίτη, αν, αναπολίτη Μισό κιλό την ημέρα δηλαδή Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται με την παραγωγή της ενέργειας που απαιτείται για την ανακύκλωση εφόσον μπορεί να παραχθεί από τα απόβλητα αυτά. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι χρειάζεται μια συνολική ολιστική αντιμετώπιση και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στις πολιτικές μας και η συζήτηση που κάνουμε σήμερα είναι τμήμα αυτών των συνολικών πολιτικών γιατί και εγώ συμφωνώ με πολλά από αυτά τα οποία λέτε. Ε, there. Λοιπόν, για τον κύριο Λαβία, εκεί στο 24 είπατε, για τον προπολογισμό. Νομίζω τα εξήγησα με σαφήνεια και το τι πιστεύω. Δεν είναι ξεκάθαρη η συζήτηση βέβαια ακριβώ τώρα. Απλά θέλω να καταλάβετε το εξής. Νομίζω ότι για τη χρηματοδότηση θα έχουμε πολύ έντονες συζητήσεις. Αλλά το πρασίνισμα της ΚΑΠ, κατά την άποψή μου, είναι ισχυρό επιχείρημα για να είναι και ικανός ο προϋπολογισμός Και αυτό είναι ένα επιχείρημα, κατά την άποψή μου, το οποίο θα αποβεί προς όφελό σας, διότι η αποδοχή εκ μέρους της κοινή γνώμης μια συνολικής περιβαλλοντικής πολιτικής είναι αρκετά υψηλή. Ρέιμερς, συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Τεχνολογία, εκπαίδευση, δεδομένα είναι τρεις μαγικές λέξεις. Και ναι, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, διότι κάποιες φορές υποτιμούμε τις απώλειες που έχουμε, γιατί δεν έχουμε τις γνώσεις σε ένα επαρκές επίπεδο. Βιοκαύσμα ήταν το επόμενο ερώτημα. Όπως ξέρετε, Κυρία Σάρμπο, ναι. Αλλά και άλλοι νομίζω με ρώτησαν πριν από την κυρία Σάρμπο. Λοιπόν, τα βιοκαύσιμα. Δεν μπορώ να σας πω δεν έχουμε στόχους, γιατί έχουμε στόχους. Στην προηγούμενη επιτροπή που συζητούσαμε το θέμα, εγώ πάντοτε υποστήριζα στεναρά να έχουμε καύσιμα δεύτερης και τρίτης γενιάς, γιατί η πρώτη γενιά ε, πρέπει να προσέχουμε. Και η βιωσιμότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα, για τα βιοκαύσιμα. Πώς θα συνεχίσουμε λοιπόν τώρα. Νομίζω το 2012 πρέπει να κάνουμε την ε, αναθεώρηση στην Κομισιόν, να δούμε πού βρισκόμαστε και να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Δεν ξέρω ακριβώς τι έκβαση θα υπάρξει, αλλά η προσέγγιση στα βιοκαύσιμα κατ' είναι μέσω της λογικής ε, οριζόντια βιωσιμότητα που θα αντισταθμίζει τις πιθανές επιπτώσεις και έτσι θα αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε. Πιστεύω ότι τα βιοκαύσιμα θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον, αλλά όπως σας είπα η βιωσιμότητα είναι το κριτήριο. Νομίζω έχω απαντήσει κατά βάση στον κύριο Νταντά εμέσως απάντησα Πιστεύω ότι έχουμε πραγματικά καλές πιθανότητες να καταλήξουμε σε κάτι που θα είναι και προς δικό σας όφελος αλλά και προς δικό μου όφελος. Σας τίνω λοιπόν χείρα συνεργασίας και ελπίζω να τη δεχτείτε. Ευχαριστώ αγαπητέ επίτροπε. Όχι μόνο ευχαριστώ για τα λόγια σου τα καλά, αλλά και για τον τρόπο που είπες αυτό που είπες και για την ευαισθησία που επιδεικνύει στον τομέα της γεωργίας. Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι περίπλοκες, απαιτούν ειδικέ προσπάθειες από πλευρά όλων. Σε ευχαριστώ λοιπόν που ήρθες ανάμεσά μας σήμερα στην Επιτροπή Γεωργίας για να μεταφέρεις τις απόψεις σου. Απόψεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές να πω επίσης ότι εμείς θα ξεκινήσουμε μία, μία έκθεση πρωτοβουλίας για... Con questo τον τρόπο με τον οποίο υπερβάλλουμε στην κατανάλωση των τροφίμων και έτσι χάνουμε μεγάλες ποσότητες. Σας ευχαριστώ όλους. Μικρή διακοπή λοιπόν.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 συνεχίσουμε λοιπόν με τα σημεία 4 και 5 της ημερησία διάταξη Θα τα εξετάσουμε από κοινού ασφαλώ σε ό,τι αφορά τα, σύστημα, τα συστήματα ποιότητα που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα. Ε, η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών έχει οριστεί για τις 3 Μαΐου. Η συγγήτρια είναι η Ράτσε Γκαρσία Πέρες που θα μας παρουσιάσει δύο νομοθετικέ ε, προτάσεις που υπάγονται σε ένα πακέτο. Πρόκειται για ένα πιο, ένα πιο σημαντικά πακέτα της Επιτροπής μας για το νέο νομοθετικό πλαίσιο της συνθήκης. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να αποστείλουμε ένα γυρό αλλά και στην ε, ε μήνυμα για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Η συγκίτρια Καρσία Περές Ε, έχει επεξεργαστεί πολλά στοιχεία σε ό,τι αφορά και την νομοθετική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να της δώσω κατευθείαν λοιπόν το λόγο, να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρευρίσκονται εδώ, τον κύριο Μαρίνο και τον άλλο συνάδελφο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συζήτηση προθεσμία για τις τροπολογίες 3η ε, Μαΐου στις 12 η ώρα. 20 Ιουνίου η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε στην Επιτροπή μας τη συζήτηση για το λεγόμενο πακέτο ποιότητας Ήδη είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία που θα έχουμε να συζητήσουμε σε σχέση και με το σχέδιο έκθεσης που έχω εκπονήσει. Όπως έχουμε προείπει, να επαναλάβω ότι θεωρώ ότι η πρόταση της Κομισιόν που έχει ως στόχο την ενίσχυση για την απλούστευση του υφιστάμενου συστήματος ε, και έχει λάβει υπόψη τη και πολλά από τα στοιχεία του Κοινοβουλίου μέσω της έκθεσης ΚΟΤΑ, αλλά παρόλα αυτά θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποια άλλα ζητήματα που δεν έχουν συμπεριληφθεί, αλλά θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Κατά την εκπόνηση της έκθεσης ε, είχαμε διάφορες συναντήσεις με την Κομισιόν, με το Συμβούλιο και με τον κλάδο γιατί στόχος μας ήταν να κάνουμε μια ισορροπημένη πρόταση, ξέροντας ότι βασικός στόχος είναι η ενίσχυση του συστήματος ποιότητας, αλλά έχοντας υπόψη ότι θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και κάποια ζητήματα τα οποία δεν είχε συμπεριλάβει η Κομισιόν στην αρχική της πρόταση. Η έκθεση λοιπόν που σας προτείνω σήμερα πρέπει να περιλαμβάνει την απλούστευση, την ανάπτυξη των υφιστάμενων συστημάτων και την πρόσθεση νέων όρων ποιότητας που μπορούν να αποτελέσουν προστιθέμενη αξία σε σχέση με τα καλύτερα ευρωπαϊκά προϊόντα. Όλοι συμφωνούμε ότι τα πρότυπα για την ποιότητα, για την ευημερία, τα οποία έχουμε ανα, ε, επιβάλει, αν θέλετε, στους Ευρωπαίους αγρότες και κτηνοτρόφους, αποτελούν προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Και αυτή η γενική σκέψη πρέπει να διέπει όλες τις προτάσεις μας για την προώθηση των ευρωπαϊκών προϊόντων και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η ποιότητα των προϊόντων μας, όπως, λέω, όπως είπα, είναι προστιθέμενη αξία που πρέπει να στηρίξουμε και να προωθήσουμε. Και πρέπει να το λέει και η σχετική νομοθεσία αυτό. Τώρα, σε σχέση με τις ε, τροπολογίες που βάλαμε για την πρόταση της Κομισιόν, θα αναφερθώ αποκλειστικά και μόνο στις ε, κατεμέ σημαντικότερες τροπολογίες. Τις έχουμε συζητήσει άλλωστε και πιο πριν στην Επιτροπή μας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν ε, κάποιες ιδιαιτερότητες. Θέλουμε να αναφέρονται στα μη ταπημένα προϊόντα. Υπάρχουν κάποιες παραδοσιακές ε, μέθοδοι παραγωγή στη γεωργία και στην κτηνοτροφία που δεν περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια και δίνουν ως αποτέλεσμα προϊόντα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ε, αποτελούν μια προστιθέμενη αξία λόγω και των γεωργικών πρακτικών. Και νομίζω ότι μπορούν να εμπέσουν στο πεδίο αρμοδιότητα αυτή τη πρόταση. Θέλουμε λοιπόν τα μη μεταποιημένα προϊόντα να συμπεριληφθούν σε ό,τι αφορά τώρα το δεύτερο τίτλο, σε σχέση με το άρθρο 5, συμφωνούμε με τους ορισμούς. Προτείνουμε πάντως να συμπεριληφθεί και ένας ορισμός του σταδίου παραγωγής για να μην υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες που θα μπορούσαν να προκύψουν αν δεν μπει αυτή η έννοια του σταδίου παραγωγής. Σε σχέση τώρα με το άρθρο 12, παράγραφος 3, ο κοινοτικό λογότυπος θεωρούμε ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικό μόνο για τα κοινοτικά προϊόντα. Και επειδή συμπεριλαμβάνεται και ήδη η προστατευόμενη ονομασία προέλευση ή γεωγραφική ένδειξη, θα μπορούσε αυτή η ένδειξη και οι συντομογραφίε προαιρετικά να αναφέρονται, να συμπεριληφθούν. Εμείς λέμε όμως να είναι υποχρεωτικό αυτό γιατί Νομίζω ότι ενισχύει ακόμη περισσότερο την ενημέρωση, την πληροφόρηση που δίνουμε στον Ευρωπαίο καταναλωτή και όχι μόνο τον Ευρωπαίο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε επίσης ότι τον κοινοτικό λογότυπο θα μπορούσαν να τον αναφέρουν μόνο όσες ονομασίες έχουν συμπεριληφθεί στο Μητρό υπό ταυτόσιμους όρους. Σε σχέση τώρα με το τέταρτο τίτλο, Ζητούμε στην ενία ΚΟΑ να συμπεριληφθούν ε, νέοι, ε, νέες προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας, προϊόν, ε, ορεινής γεωργίας, παραδείγματος χάρη, αυτόχθονο προ κτλ. Επίσης θα πρέπει να έχουμε και ένα σύστημα για την επισήμανση των προϊόντων από βοηδή. Για την ορεινή γεωργία το έχουμε ξαναπεί και στην έκθεση Σκότα ήταν ε, μεγάλη η πλειοψηφία που υποστήριξε τη συμπερίληψη και θέλαμε λοιπόν και εμείς να το αναφέρουμε για να συμπεριλαμβάνεται και στον κανονισμό για το σύστημα ποιότητας. Σε ό,τι αφορά και τις ΠΟΠ και τις ΠΓΕ, ε, θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε στον κανονισμό αυτό ποιότητα, στο σύστημα ποιότητας ε, τις γεωγραφικές, τις ε, προστατευόμενε ονομασίες προέλευσης και προστατευόμενε γεωγραφικέ ενδείξεις, αλλά και κάποιε προαιρετικέ ενδείξει, Παραδείγματο χάρη όπως είπα προϊόν ορεινή γεωργίας. Αλλά πρέπει και οι προαιρετικέ ενδείξει νομίζουμε να περάσουν στην ενιαία ΚΟΑ. Αυτές οι προαιρετικές ενδείξεις είναι κάτι διαφορετικό από τις προστατευόμενες ονομασίες ε, προέλευση και γραφικές ενδείξεις. Τώρα, στον τίτλο 5 θα θέλαμε να υπάρξει μια παράγραφος για τη χρήση των συστατικών. Η Κομισιό νομίζουμε ότι πρέπει να κάνει μια σχετική μελέτη. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε και το θέμα αυτό. Ένα άλλο στοιχείο που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό και το ζητά και ο κλάδος. Και φαντάζομαι θα το στηρίξουν και πολλοί συνάδελφοι. Είναι ο ρόλος των ενώσεων παραγωγών. Πρέπει να υπάρχουν εργαλεία που θα δίνουν τη δυνατότητα σε ομάδες παραγωγών να έχουν ένα ρόλο για ε, ε, για την παραγωγή. Έχουμε το άρθρο 48.3 και εκεί προτείνουμε να γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις ε, για την επίτευξη συμφωνίας και σε ό,τι αφορά τις ομάδες παραγωγών, τις ενός παραγωγών, να εξηγήσω έτσι λίγο πιο λεπτομεριακά, γιατί το συζητούμε πολλές φορές, το συζητούμε και με τις οργανώσεις παραγωγών στις χώρες μας, υπάρχει μια τροπολογία που λέμε ότι σε ό,τι αφορά αυτό το σύστημα, αυτά τα συστήματα διαχείρισης προσφοράς δεν θα πρέπει να πλήξουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά, ούτε να αποτελέσουν εμπόδιο για νέους φορείς στην αγορά ούτε να πλήξουν αρνητικά τους μικρούς παραγωγούς. Θα υπάρχει σχετική κοινοποίηση στην Κομισιόν, η οποία θα μπορεί να ανακαλεί ανα πάσα χρονική στιγμή κτλ. Δηλαδή, τι λέμε, είναι σημαντικό οι οργανώσεις, οι ενώσεις των παραγωγών να μπορούν να έχουν στα χέρια τους κάποιο είδους εργαλείο για τον έλεγχο των όγκων, όπως λέμε, των ποσοτήτων, αλλά με τους απαιτούμενους ελέγχους βέβαια και χωρίς αυτό να μπορεί να θίξει μικρούς παραγωγούς. Γι' αυτό λοιπόν θελήσαμε στην τροπολογία την οποία υποβάλλουμε να είναι ξεκάθαρο. Αφενός να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος των ομάδων παραγωγών για τον έλεγχο των ποσοτήτων, αλλά και σε ό,τι αφορά τους ελέγχους εκ μέρους των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν θα πρόκειται σε τέτοιους ελέγχους. Eh, Αυτά είναι λοιπόν τα σημαντικότερα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα στο πλαίσιο αυτής της πρότασης που υποβάλλουμε σε σχέση με τον κανονισμό περί συστήματος ποιότητας. Όπως είπα, συμφωνεί και με τις ανησυχίες και τις προτάσεις του κλάδου, αλλά και με τα όσα προέκυψαν και από τις συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων που είχαμε μεταξύ εδώ των συντρόφων της Επιτροπής της Επιτροπής Γεωργίας και σε ό,τι αφορά τα πρότυπα εμπορίας και τη σχετική οδηγία, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο κανονισμός αυτός είναι προέρχεται από την ανάγκη υλοποίηση τη συνθήκη τη Λισαβόνα, να υπάρχουν κάποια γενικά πρότυπα εμπορία δηλαδή, για τα προϊόντα που δεν έχουν κάποια ειδικά πρότυπα. Έχουμε κάποιους ε, αποκλειστικούς όρους, προαιρετική αποκλειστική όρη, το αναφέρουμε ξανά αυτό. Παραλαμβάνω ότι ο κλάδος ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική συνεργασία μαζί του. Μας είπαν επίσης και από την Κομισιόν ότι δεν προτίθεται ούτε να καταργήσει ε, τα πρότυπα, ούτε όμως και να τα πολλαπλασιάσει. Ελπίζουμε λοιπόν να φέρουμε σε αίσιο πέρα ε, την εξέταση των ε, προτάσεων για τον κανονισμό αυτό στο πεδίο των αρμοδιτών που έχουμε ως κοινοβούλιο. Θα ήθελα ολοκληρώνοντας να πω ότι με πολύ ενδιαφέρον θα ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων. Ευθύ εξ αρχή θελήσαμε να είναι έκθεση, η έκθεση αυτή άρτια και ισορροπημένη. Να ενισχύσουμε το σύστημα ποιότητα και να το προσαρμόσουμε στι νέε ανάγκε οι οποίε ανακύπτουν ε, συν το χρόνο. Φυσικά θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους να συνεισφέρουν και να κάνουν τις προτάσεις τους, αλλά θέλουμε ένα ισχυρό σύστημα, αγαπητοί συνάδελφοι, γι' αυτό δεν θα έπρεπε να διευρύνουμε και να επεκτείνουμε πάνω στο πεδίο εφαρμογή και, και το πεδίο πάνω στο οποίο θα θέλουμε να υπάρξουν κάποιε τροποποιήσεις. Ελπίζω με το διάλογο που θα έχω με τους συντρόφους, που θα ήθελα να είναι επικοδομητικός, να καταλήξουμε σε μια καλή πρόταση και τώρα περιμένω να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων σε σχέση με την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά εξαιρετική η δουλειά που έκανες. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Με τον κύριο Σμιτ να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, ναι, ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, δουλειά που έκανε. Νομίζω ότι όντως έτσι είναι. Κοιτάζοντας και την έκθεση, Και ακούγοντας και αυτά που μας είπε η συγγήτρια, εμείς από πλευράς του ΕΛΚ θα συμφωνήσουμε πολλά από αυτά που αναφέρετε. Και νομίζω ότι μετά από συμφωνία και με τις ομάδες και με τους συναδέλφους ε, θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια κάποια στοιχεία. Να αναφέρω τα πιο σημαντικά στοιχεία, τα περί Νομίζω ότι αυτό μας βρίσκει σύμφωνους όλους εδώ στο Κοινοβούλιο. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η προσέγγιση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μείωση των προθεσμιών. Σε ό,τι αφορά και τη συμφωνία μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί είναι αρκετά οδυνηρή στην παρούσα φάση η διαδικασία και πολλές ε, ε, σε πολλές περιπτώσεις διαρκούν χρόνια οι διαδικασίες αναγνώρισης. Και υπάρχουν κράτη τα οποία είναι κατά τέτοιων περιγραφών, τέτοιων επωνυμιών και ε, αυτό καθυστερεί. Το βασικό ζήτημα είναι το εξής. Το είπε και η Ευρωπαϊκή και η εισηγήτρια, το πώς μπορούμε να ελέγξουμε την ε, ζήτηση και ποιος είναι ο ρόλος των ε, ενώσεων μελωτών. Αυτό που είναι σαφές είναι το εξής. Ότι μπορεί να υπάρξει έλεγχος της ε, ζήτησης, αλλά αυτό δεν μπορεί να θέσει σε αμφισβήτηση τον δημόσιο χαρακτήρα της επιγραφής. Δεν είναι ιδιωτικό, ιδιωτικό αγαθό ενός ομίλου, για παράδειγμα, μια τέτοια επωνυμία, θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η εγγύηση για όλους τους παραγωγούς ε, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην επωνυμία αυτή. Αυτό νομίζω ότι είναι μια βασική αρχή. Τούτου λεχθέντος θεωρώ ότι είναι θεμελιώδου σημασίας να βρούμε μια σωστή λύση προκειμένου σε ό,τι αφορά τις ε, ε, ενώσεις και προστασίες λοιπά να μπορέσει να ελεγχθεί η ζήτηση. Γιατί στην Ευρώπη βλέπουμε ότι ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προέλευση, την ε, ονομασία προέλευσης, όπου και το πώς παράγεται ένα προϊόν, εμ, οδηγεί στην εξή κατάσταση. Ο ιδιωτικός παραγωγός ε, καταλήγει να έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Σε σύγκριση με τον καταναλωτή, για παράδειγμα, όταν λέμε παρμεζάνα ρετζάνο, το πάρμα, στις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες ιδιαίτερα που το εκμεταλλεύονται αυτό, ε, μειώνονται οι τιμές και νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί η θέση των ε, ενώσεων προστασίας καταναλωτή και σύμφωνο σε ό,τι αφορά τις ορεινές περιοχές να υπάρξει πιο έντονη υποστήριξη σωστή η προσέγγιση της ηγήτριας αυτό που είναι σημαντικό θεωρώ είναι να προστατεύσουμε την επωνυμία ορεινή περιοχή, να δημιουργήσουμε μία αναφορά σε ορεινές περιοχές προκειμένου να μην υπάρχει δυνατότητα το γάλα ή το τυρί των ορεινών ε, περιοχών να αναφέρεται μάλλον ορεινή περιοχή ενώ δεν πληρούνται οι κατάλληλοι όροι, τα κατάλληλα κριτήρια. Θα πρέπει αν ένα προϊόν αναφέρει την ε, λέξη ορεινή περιοχή, να προέρχεται όντως από ορεινές περιοχές. Να πω επίσης ότι η προστασία των επωνυμιών ε, σε διεθνές επίπεδο είναι πολύ ε, πιο αδύναμη από ότι οι ιδιωτικές επωνυμίες, δυστυχώς τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και κυρίως στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κλείνοντας, σε ό,τι αφορά την, ε, τα παραδοσιακά προϊόντα, τα μη μεταποιημένα. Για τα μη μεταποιημένα λοιπόν προϊόντα, είμαι επί της αρχής υπέρ, να είναι σαφές για ποια προϊόντα ενδιαφερόμαστε. Υπάρχουν τέτοια προϊόντα στην αγορά όπου η επωνυμία αυτή θα ήταν ε, απαραίτητη. Νοπά προϊόντα, μη μεταποιημένα προϊόντα. Νομίζω ότι αν υπάρχουν τέτοια προϊόντα θα πρέπει να επιτρέψουμε αυτή την περιγραφή. Ευχαριστώ τον κύριο Ντόρφμαν για μια σημαντική παρέμβαση. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω το Συμβούλιο. Έχουμε τον πρόεδρο της ειδική Επιτροπής Γεωργίας, τον κύριο Βάιντερ, από την Ουγγρική Προεδρία και τον ευχαριστώ για την παρουσία του. Ο κύριο Σμιτ. Θα είμαι σύντομος. Υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία συμφωνούμε. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και πολύ καιρό και το θέμα της ποιότητας γενικά είναι σημαντικό. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια και να θέσω ορισμένες ερωτήσεις. Σχετικά με τη διαχείριση της προσφοράς και τον ρόλο που μπορεί να παίξει. Φοβάμαι ότι υπάρχει ανεπαρκής ευελιξία στους εθνικούς κανόνες, όποιοι και αν είναι αυτοί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινδυνεύει με την παρέμβασή της να οδηγήσει σε περίπλοκα συστήματα τα οποία δεν θα αφολήσουν. Για τα ορεινά προϊόντα είμαστε όλοι σύμφωνοι, πρέπει να είναι σε μια ειδική κατηγορία και πρέπει να την χάνουν τις ίδιες αντιμετώπισης ε, μεταξύ τους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δει κατεπηγόντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα μη επεξεργασμένα προϊόντα στα πλαίσια του καθεστώτος TSG. Δεν υποστηρίζουμε τόσο την τροπολογία 37 σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις μετά από τριετή λειτουργία. Νομίζω ότι ένα από τα ωφέλη του συστήματος ακριβώς είναι ο ανεπίσημος χαρακτήρας και το να ζητάει κανείς να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση μέσα σε μια τριετία είναι υπερβολικό. για τις άμεσες πωλήσει. Το θέμα της ετικετοθεσίας τίθεται. Δεν υπήρχε εξ αρχής στην πρόταση της Επιτροπής και πρέπει να επανεξεταστεί. Προέρχομαι από τη Σκοτία και ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα έτσι ώστε η, ο όρος ονομασίας προέλευσης να είναι σαφέστατα γεωγραφικός, γιατί κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες ακολουθούν άλλες λογικές. Νομίζω ότι γενικά η κατεύθυνση της πρότασης είναι σωστή και στα πλαίσια της συνάντησης των σκιωδών εισηγητών, στην επόμενη που θα έχουμε, θα συνεργαστούμε σωστά. Ρέινερτς και μετά Σκοτά. Σας ευχαριστώ. Πολλά ήδη ακούσαμε. Αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι το εξής. Αν υπάρξουν ρυθμίσεις, ε, να παραμένουν εθελούσιες γιατί υπάρχει γεωγραφική προέλευση, ονομασία προέλευσης και αν αυτό καταστεί αυτό υποχρεωτικό χάνεται ένα πλεονέκτημα για τον ε, παραγωγό γιατί δεν υπάρχει πλέον διάκριση και δεν μπορεί κανείς να διακριθεί από τους υπόλοιπους παραγωγούς της ε, περιοχής τους. Αυτό που μας κάνει επίσης εντύπωση είναι ο λογότυπος, το ευρωπαϊκός λογότυπος και οι τρεις λογότυποι ουσιαστικά δεν είναι γνωστοί στους πολίτες, δεν είναι αναγνωρίσιμοι. Και ίσως θα μπορούσαμε να συνδέσουμε την επωνυμία με το λιγότυπο για να υπάρξει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα. Γιατί αν δεν καταφέρουμε να καταστούν γνωστά, γνωστοί αυτοί οι λογότυποι, δεν έχει νόημα να υπάρχει αυτή η σφραγίδα γιατί δεν υπάρχουν πλέον τα εμπορικά πλεονεκτήματα. Άρα θεωρώ ότι η σύνδεση λογότυπου και επωνυμίας είναι πιο σωστή από το να αναφέρεται ένα από τα δύο μόνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρώ τη συνάδελφο για την έκθεσή της η οποία είναι πολύ καλή. Χαίρομαι επίσης γιατί οι προτάσεις οι οποίες έγιναν σε επίπεδο εισηγητών σκιωδών έγιναν δεκτές, ιδιαίτερα για την ορεινή παραγωγή. Το ειδικό αυτό καθεστώς είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για να υπογραμμιστεί προς τον καταναλωτή η προστιθέμενη αξία των ορεινών προϊόντων, αλλά γιατί βοηθά αυτές τις ορεινές περιοχές, οι οποίες είναι λιγότερο ευνοημένες, εισαγωγικά για το ποιοτικό καθεστώς των παραδοσιακών σπεσιαλιτέ. Νομίζω ότι και εδώ ωφελούμε κάποιες ομάδες παραγωγών δημιουργώντας τους τη δυνατότητα δημιουργίας καθεστώτος σωστών, σωστής διαχείρισης του προϊόντος. Υπάρχουν κάποια προβλήματα σχετικά με την νομική εγγύηση η οποία θα πρέπει να παρέχεται στις ονομασίες προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 42. Τώρα σχετικά με τους ε, κανόνες με τους οποίους ε, οι ονομασίες αυτές προέλευσης θα μπορεί να χρησιμοποιούνται. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να υπάρξει σωστός έλεγχος, πρέπει να διευκρινιστεί. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω τον ρόλο των οργανώσεων των παραγωγών σχετικά με την προσαρμογή της ζήτησης, η οποία πολλές φορές δεν μπορεί να καλύπτεται εύκολα. Παναλαμβάνω ότι η έκθεση πάντως είναι πολύ καλή και θα συνεχίσουμε τη σωστή συνεργασία. Ευχαριστώ Τζαν Καύλο Ζωζέ Μποβέ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία στην έκθεσή της το ότι δεν υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στις διαφορετικές ονομασίες προέλευσης, το ότι σημειώνουμε ότι η προστιθέμενη αξία είναι περισσότερη από ό,τι στα λεγόμενα απλά προϊόντα και αυτός είναι λόγος αναγνώρισης, το ότι υπάρχει μια αγροοικολογική πλευρά του συστήματος ονομασίας προέλευσης, όλα αυτά είναι σημαντικά και επίσης είναι συμβατά με το διεθνές εμπόριο. Ε, βέβαια εκεί θα υπάρξουν σημαντικές συγκρούσεις και με τις Ηνωμένε Πολιτείε για το λεγόμενο trademark. Εδώ θα πρέπει να είμαστε σαφείς σε επίπεδο Ευρώπης και θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε και στο Κοινοβούλιο ότι δεν θα πρέπει να υποκύψουμε στο Συμβούλιο έτσι ώστε η έννοια ετικέτας ποιότητας να μην περιορίζεται στα ευρωπαϊκά σύνορα. Τώρα, για κάποια θέματα στα οποία διαφωνώ, θα έλεγα, με την εισηγήτρια, όταν ζητάμε μία απλοποίηση των διαδικασιών, δεν είναι κακή ιδέα, η απλοποίηση των διαδικασιών ταυτόχρονα όμως μπορεί να προκαλέσει και τη μείωση των κριτηρίων που συνιστούν τη συγκεκριμένη αυτή αναγνώριση. Εδώ απαιτείται λοιπόν μια διαδικασία αναγνώρισης πολύπλευρη και πολυεπίπεδη και αν υπεραπλουστεύσουμε τα πράγματα φοβάμαι ότι θα καταστήσουμε αδιάφορα και ουδέτερα τα συστήματα αυτά. Ένα τελευταίο σημείο με το οποίο έχω πρόβλημα είναι το θέμα των, των μονάδων εκμετάλλευσης. Υπάρχει εδώ αναγνωρίζουμε ένα πρόβλημα να γίνουν, να προσαρμοστούν προς τους κανόνες οι μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό αναγνωρίζεται στην αιτιολογική σκέψη, αλλά στο κείμενο, το νομικό, δεν υπάρχει μια τέτοια αναγνώριση. Η πρόθεση υπάρχει μεν, αλλά πρέπει να περιλαμβάνεται και στη διατύπωση. Και μετά μπορούμε να συζητήσουμε για πιο περίπλοκα θέματα όπως ε, οι εμπορικοί κανόνες, όπου ισχύει ένα σύστημα το οποίο βασίζεται θα έλεγα στα βιομηχανικά προϊόντα και δεν λαμβάνει υπόψη την διαφορετικότητα των τρόπων παραγωγής. Αν εμείς ε, διακανονίσουμε θα έλεγα σε επίπεδο ευρωπαϊκό μόνο τότε θα περιθωριοποιήσουμε ορισμένα προϊόντα τα οποία ε, δυστυχώς δεν θα συμπεριληφθούν με αυτόν τον τρόπο. Κατά τα άλλα η έκθεση είναι εξαιρετική. Ευχαριστώ Νταντέν και μετά Μάτω. Ευχαριστώ. Θέλω καταρχάς ε, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και για τη δουλειά που έκανε και γιατί έλαβε υπόψη τι απόψεις των πιο ενδιαφερομένων ε, μέλων της Επιτροπής μας για το θέμα. Θα ήθελα να αναφέρω ένα θέμα για την ποιότητα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να προσθέσουμε κάτι σε ό,τι αφορά την πιθανή συνεργασία μεταξύ κρατών και κομισιών, αν υπάρξει κάποια σφετερισμός ή ε, κάποια σήματα ποιότητας, ε, ε, υπάρξει κάποια κατάχρηση. Διότι υπάρχει ε, δυσκολία σήμερα. Δεν μπορούμε ποινικά να αντιμετωπίσουμε τέτοια κρούσματα με εύκολο τρόπο. Τώρα επανέρχομαι στο δεύτερο κείμενο, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα πρότυπα εμπορία. Νομίζω ότι μέσα από τις γραμμές υπάρχουν κάποια επικίνδυνα στοιχεία που ουσιαστικά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με αυτά τα οποία προασπίζουμε εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια στην Επιτροπή μας. Από το σχέδιο κειμένου προκύπτει ότι έχουμε τρία σημεία των οποίων ε, η πρόταση αυτή δεν φαίνεται να είναι ε, συνεπής. Παραδείγματος χάρη με το μοντέλο Γεωργίας που μιλά για τον για το σεβασμό των διεθνών ε, διατάξεων, ότι παραδείγματο χάρη λέει ότι υπάρχουν κάποιες απαιτήσει υψηλότερε σε ό,τι αφορά τα ζωικά προϊόντα σε σχέση με τον κόντεξ αλιμεντάριους για να ανταποκριθούμε στι προσδοκίε του Ευρωπαίου καταναλωτή, που πολλέ φορέ λέμε δεν είναι προσδοκίε ε, των καταναλωτών από άλλε υπήρου. Αν εφαρμόσουμε το κείμενο ω έχει, αυτό σημαίνει ότι αύριο θα μπορούσαν αυτά τα προϊόντα να μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ίσως θα μπορούσαν να καταπέσουν όλες οι ρυθμιστικές διατάξεις που είναι αυστηρότερες και που έχουν εφαρμοστεί για κάποια προϊόντα. Και αυτό θα έχει και να κάνει και με κάποια προϊόντα ποιότητα για το οποίο θέλουμε να υπάρχει σήμα Και τελευταίο, μιλάμε για την ποιότητα, αλλά δεν ορίζεται ξεκάθαρα και έτσι θα υπάρξουν δυσκολίες για τον έλεγχο και από τους ίδιους παράγοντες αλλά και από τις επίσημες ε, υπηρεσίες ελέγχου. Άρα θα πρέπει με τροπολογίες να διευκρινίσουμε τι εννοούμε ακριβώς ποιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Μάτο και μετά είναι προφανές ότι στην πολιτική ε, ποιότητα με τον νέο επίτροπο είχαμε μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τη θέση που είχε ακολουθήσει η προκάτοχός του. Αυτό πρέπει να μας γεμίζει ικανοποίηση. Η πρόταση της ε, Κομισιόν γενικά είναι καλή. Σημαντικό ήταν αυτές οι ονομασίες ε, προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη να διαχωριστούν. Αυτό θέλαμε και το πετύχαμε. Επίσης, το να υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας ονομασιών με μια πρώτη και μια δεύτερη ονομασία και αυτό δεν έγινε δεκτό. Τώρα σε ό,τι αφορά την έκθεση της συγκεκριτρίας νομίζω ότι αξίζει χαρητηρίων. Είναι μια πάρα πολύ καλή έκθεση η οποία ανταποκρίνεται και στις ανησυχίες των παραγωγών αλλά και της ισπανικής αντιπροσωπείας ε, του Λαϊκού Κόμματος. Εμείς πιστεύουμε και θέλω να τονίσω το εξή ότι η επανεισαγωγή στον ορισμό των ονομασιών προέλευσης και της μεταποίησης και της προετοιμασίας από συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή είναι κάτι σημαντικό, είναι και ένα σημαντικό επίτευγμα σε σχέση με την αρχική πρόταση. Και βέβαια η αναφορά στα προϊόντα ορεινής γεωργίας είναι σημαντικό και θα ήθελα να μιλήσω και για τα αυτόχθονα αυτά προϊόντα που επίσης είναι πολύ σημαντικό. Τώρα κάτι άλλο. Να δυνατότητα κατάργησης του να μπορούν προϊόντα τρίτων χωρών να χρησιμοποιούν τα σύμβολα και τις ενδείξεις τις κοινοτικέ. Ίσως και η συγκήτρια να προσπαθεί να υπάρξει μεγαλύτερος έλεγχος, αλλά είναι κάτι το οποίο επανέρχεται συνέχεια, μας ανησυχεί και εμείς σίγουρα θα καταθέσουμε σχετική τροπολογία. Τέλος, κάτι άλλο που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι πάλι δεν έχουμε την εισαγωγή ενός ειδικού καθεστώτος ε, γεωργίας για την ολοκληρωμένη παραγωγή. Αυτό το ζητά ο κλάδος εδώ και πολύ καιρό και αυτό μπορεί να δώσει για αξία στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Και σε ό,τι αφορά τα πρότυπα εμπορία τώρα, να θέσω το εξή. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι για το μέλλον προτίθεται να ενισχύσει τα πρότυπα εμπορίας αλλά η προβλεπόμενη δικασία στις κατεξουσιοδότηση πράξης θα μπορούσε να είναι δίκοπο μαχαίρι. Και είχαμε τη σχετική εμπειρία ήδη σε σχέση με τον τομέα των κυπευτικών. Ούτε ενισχύθηκε, θα έλεγα ότι και αποδυναμώθηκε ο τομέας. Επομένως το αφήνω αυτό έτσι, να πλανάται ως προειδοποίηση και πρέπει να το προσέξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Molto bene, grazie onorevole Mato. Stefan James Nicholson. Stefan τώρα και μετά James Nicholson. Και εγώ θέλω να συγχαρώ με τη σειρά μου την εισηγήτρια για την έκθεση που μας προτείνει. Συμφωνώ με πολλά από όσα είπε για τα αριθμιστικά κυρίως ο Μισελ Νταντά, να τονίσω όμως δύο πράγματα. Πρώτον, το διεθνές επίπεδο, ότι πρέπει να επιμείνουμε, ιδίως απέναντι στην Κομισιόν, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων να προσπίσουμε τα δικά μας συμφέροντα και να επανεπιβεβαιώσουμε ξεκάθαρο ότι η ποιότητα ανήκει και εντάσσεται πλήρως στην Ευρω... στρατηγική της Ευρώπης. Έχουμε μια μισή φορά παραπάνω ε, προστιθέμενη αξία από τη ΣΥΠΑ. Μια μισή φορά παραπάνω λοιπόν στα οποροκρευτικά γενικά στα βαρβατικά προϊόντα. Αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε. Και αυτό το οποίο προτείνεται για τις ομάδες παραγωγών, γιατί το σήμα πάει χέρι με χέρι με μια ομάδα παραγωγών. Πρέπει να το έχουμε υπόψη αυτό. Θα πρέπει να το σκεφτούμε λοιπόν πολύ προσεκτικά, γιατί όταν έχουμε παραγωγή ποιότητας, τη ζήτηση δεν την καθορίζει μόνο η αγορά και η προσαρμογή είναι δύσκολη μεταξύ των μεταποιημένων ποιοτικών προϊόντων και του εποπόδου και του όγκου παραγωγής. Πρέπει εκεί να υπάρχει μια ομάδα, μια οργάνωση παραγωγών η οποία θα πρέπει να συγκροτηθεί και να διαχειρίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα αυτά τα θέματα. Πρέπει να τα σκεφτούμε λοιπόν και αυτά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη γραμμή και αυτό θα προσπαθήσω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, James Nicholson και Μάριν Μαγκίνες στη συνέχεια. you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα να καλωσορίσω την έκθεση της εισηγητριάς και να τη συγχαρώ ασφαλώς για την έκθεση αυτή. θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να μην περιπλέξουμε την κατάσταση πιο πολύ από ό,τι χρειάζεται. Θα πρέπει να δούμε μία από τις μεγάλες λύσεις ε, για την κατάσταση, γιατί αν και ο καταναλωτής, αν και τον καταναλωτή τον ε, βομβαρδίσουμε με πληροφορίες, δεν θα μπορέσει να τις απορροφήσει όλες. Η προέλευση αποτέλεσε εδώ και καιρό ένα πρόβλημα, το οποίο συζητιέται πολύ έντονα στην Επιτροπή μας από πολλές απόψεις. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί προκειμένου να μην επιβαρύνουμε υπερβολικά. Προτεραιότητα θα πρέπει να είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Τα προκυπευτικά που θα έρχονται εκτός Ένωσης θα πρέπει καταρχάς να διευκρινιστεί ότι δεν ε, ε, έχουν παραχθεί στην Ένωση και μιλάω και για τα πουλερικά και για το κρέας ε, σε χώρες που έχουν παραχθεί σε χώρες του Μερκοσούρ. Άκουσα με ενδιαφέρον και καταλαβαίνω τα προβλήματα που τονίζουν οι συνάδελφοι και νομίζω ότι αποτελούν ε, από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η Επιτροπή μας για το μέλλον, γιατί πολλές από τις αποφάσεις που παίρνουμε τώρα, ακόμα και όταν κινούμαστε από την έκθεσή μου, για παράδειγμα, στο γάλα, για το γάλα, για ποσοστώσεις απειλούμε ίσως και διακυβεύεται το μέλλον όσων ε, δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό γιατί επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητά τους. Και ασφαλώς ε, τα PDI μπορεί να είναι ένας τρόπος να προστατεύσουμε κάποιες ε, συγκεκριμένες περιοχές. Νομίζω ότι από πλευρά μου κάτι που μας έχουν διδάξει οι εμπειρίες των τελευταίων δέκα ετών είναι θα πρέπει να έχουμε τα υψηλότερα πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το θέλει ο καταναλωτής. Θέλει να ελέγχεται η παραγωγή των τροφίμων με υψηλά πρότυπα. Αλλά πρέπει να πω, ακούγοντας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν μιλούν για τα προκυπευτικά εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το να πληρούν τα ίδια πρότυπα. Μιλούν για παρόμοια πρότυπα. Συγγνώμη, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των ιδίων προτύπων και παρόμοιων προτύπων. Αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε επίσης. Να καταστήσουμε σαφές ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε να περάσουν παρόμοια πρότυπα, κάτω από τα δικά μας πρότυπα δηλαδή. Grazie James, chiude McGuinness. Μαγκίνες θα κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή, την εισηγήτρια μάλλον. Το θέμα είναι πώς συνδυάζονται αυτά που είπατε με την ομοθεσία για την ενημέρωση του καταναλωτή σε σχέση με την προέλευση των προϊόντων. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα ψηφίσει το Κοινοβούλιο στον τομέα της ονομασίας προέλευσης και πώς αυτό θα επηρεάσει τις διαφορετικές ρυθμίσεις οι οποίες ισχύουν στις διάφορες χώρες. Το δεύτερο ότι διάφορες χώρες λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Χαίρομαι βέβαια που τα πράγματα τα αντιμετωπίζουμε με μια κάποια όρεξη σήμερα επειδή είναι Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας, αλλά υπάρχουν τεράστια εμπόδια για πολλούς από τους συναδέλφους και δεν ξέρω ποιοι είναι οι ορισμοί για τις ορεινές περιοχές οι οποίοι να ταιριάζουν θα έλεγα για το μεγάλο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι για τοπικές περιπτώσεις μόνο. Θα ήθελα λοιπόν κάποιες διευκρινήσεις επιγόντως σε σχέση με αυτό. Ευχαριστώ κύριε Μαγκίνες. Θα δώσω τώρα το λόγο στην υποδιευθύντρια της ειδική Επιτροπής και μετά στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε το ότι η προάσπιση της ποιότητας περνάει μέσα από έναν ρόλο τον οποίο παίζουν οι οργανώσεις που ελέγχουν και συνοδεύουν τα προϊόντα και μπορούν να επηρεάσουν και τον προγραμματισμό της παραγωγής και αυτό είναι ποιοτικό χαρακτηριστικό και όχι μόνο χαρακτηριστικό ενίσχυσης της εμπορίας. Για την ετικετοθεσία νομίζω ότι όπως είπε και η Μαγκίνες θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτά τα οποία είπε ήδη η Επιτροπή μας σχετικά με τις ρυθμίσεις για την ενημέρωση του καταναλωτή. Νομίζω ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε θετικά για τους ενδιαφερομένους πάντως. Λορέτα Μαρίνο πρώτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πλήρη έκθεσή της να ευχαριστήσω για την υποδοχή που έτυχε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαπιστώνω με χαρά ότι υπάρχει κοινό στόχος ότι σε ενίσχυση των συστημάτων ελέγχου της ποιότητας και για τον παραγωγό και για τον καταναλωτή. Θα αναφερθώ στις ίδιες τροπολογίες, τις οποίες αναφέρθηκε η συγγήτρια και να προσπαθήσω να εξηγήσω τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάπως καλύτερα. Πρώτον, το ότι διευρύνουμε τις παραδοσιακές αυτές, τα παραδοσιακά προϊόντα και στα μη επεξεργασμένα προϊόντα. Η προσπάθειά μας είναι να διευκρινίσουμε αυτά τα προϊόντα καθιστώντας τα πιο συγκεκριμένα και διαφοροποιώντας τα από τα άλλα συστήματα έτσι ώστε ο καταναλωτής, ο οποίος έχει ήδη κάποιες δυσκολίες να διακρίνει τις διαφορετικές ετικέτες, να μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να προσανατολιστεί σωστά. Αυτός είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάμεσα σε άλλους βέβαια, ε, στη μείωση ε, των προϊόντων αυτών στα μη επεξεργασμένα προϊόντα. Σχετικά τώρα με τις δυσκολίες ε, για τον καθορισμό των φάσεων της παραγωγής, λαμβάνουμε υπόψη την ανάγκη που υπάρχει στον τομέα αυτό. Αυτά τα οποία προτείνονται στην έκθεση σε σχέση με αυτό δεν λύνουν το πρόβλημα. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν τα πράγματα καλύτερα έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι φάσεις της παραγωγής για την αναφορά στο άρθρο 12 παράγραφος 3 και στην, στον υποχρεωτικό, στην υποχρεωτική σήμανση. Λαμβάνουμε υπόψη μας αυτά που είπε η συγγήτρια, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας και σε ένα πρόβλημα, ένα μπούμεραν ουσιαστικά, σχετικά με τον περιορισμό του, της χρήσης του τόπου για ξένα προϊόντα σε προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί θα έλεγα την μεμονωμένη διαδικασία έγκρισης τύπου σαν ειδικά προϊόντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας βάλει σε δύσκολη θέση στα πλαίσια των διμερών διαπραγματεύσεων που έχουμε. Γιατί όταν έχουμε κάποιες διμερείς διαπραγματεύσεις, εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πάρα πολλά προϊόντα τα οποία θέλουμε να προασπιστούμε, από την άλλη πολλές φορές έχουμε μεμονωμένες χώρες με λίγα προϊόντα και αν εμείς περιορίσουμε τη χρήση ε, του τύπου <clears throat> σε κάποιες μόνο διαδικασίες ε, τότε θα καταστήσουμε τις διαπραγματεύσεις μας ε, με τους εταίρους μας πολύ πιο δύσκολες. Γιατί επαναλαμβάνω τα αντίστοιχα προϊόντα στις χώρες αυτές που πολλές φορές προσφέρονται προς κατάχρηση των δικών μας προϊόντων είναι προϊόντα τα οποία δεν αποφεύγουμε την πώλησή τους στις αγορές μας. Σχετικά τώρα με τους, ε, με τους όρους λειτουργίας της ενιαίας ε, αγοράς, Τη ενιαίας ΚΟΑ, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση των ειδικών χαρακτηριστικών του προϊόντος και σε ποιοτικό επίπεδο και από την άλλη έχει μεγάλη σημασία να συγκεντρώνει όλες τις ενδείξεις οι οποίες περιλαμβάνονται στα διαφορετικά νομικά μέσα που είναι στη διάθεσή μας και που έχουν ένα κομμάτι της νομικής τους βάσης στο Συμβούλιο και άλλο ένα στην Επιτροπή. Αυτό θα προσδώσει συνεκτικότητα στο σύστημα. Ειδικά τώρα με αυτά τα οποία λέγει η συγγήτρια στην έκθεση που ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κατευθυντήριες γραμμές της γύρω από τη χρήση των συστημάτων αυτών στα μετασχηματισμένα προϊόντα και σχετικά με τα ιδιωτικά συστήματα πιστοποίησης θα λάβουμε υπόψη μας το συγκεκριμένο αίτημα. γύρω από το θέμα της οργάνωσης των παραγωγών, των οργανώσεων των παραγωγών. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ είναι σχετικά επιφυλακτική. Εμείς θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο κανονισμός αναγνωρίζει το ρόλο των οργανώσεων των παραγωγών. Μέχρι τώρα μια τέτοια αναγνώριση είχε γίνει αντικείμενο αναγνώρισης μόνο για την διαδικασία καταγραφής του προϊόντος. Αναγνωρίζουμε το ρόλο τους λοιπόν και στον τομέα της εγγύησης της ποιότητας και της παρακολούθησης της αγοράς και της ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών σε περίπτωση προβλήματος. Μια πιο επιφυλακτική θέση σε σχέση με τη διαχείριση της παραγωγής. Η γεωγραφική ένδειξη προϊόντος έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με τα προϊόντα τα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται όποιος προχωρά στη διαδικασία αυτή για να εντάξει το προϊόν του δεν είναι υποχρεωμένος να ανήκει σε μια ευρύτερη ομάδα. Συνεπώς εδώ δημιουργούνται κάποιες ανησυχίες από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόταση της εισηγήτριας γύρω από τις πιθανές αντιθέσεις με την οδηγία για τον ανταγωνισμό και ιδιαίτερα ανησυχίες σχετικά με τα νέα προϊόντα. Σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν την επιφυλακτικότητα με την οποία η εισηγήτρια δέχεται την συγκεκριμένη τροπολογία στην έκθεσή της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το ενδιαφέρον που έχει η εισηγήτρια για την ε, τροπολογία της σχετική με την εισαγωγή της ε, ε, ποιοτικής ένδειξης ορεινό προϊόν ορεινής προέλευσης του προϊόντος. Αυτό δεν είναι κάτι το καινοτόμο θα έλεγα. Είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει και έχουμε ήδη εξετάσει ήδη από το 1908, από το 2008 στα πλαίσια της απάντησης που δώσαμε στην, στο πράσινο βιβλίο. Είναι κάτι το οποίο εξετάζει ακόμα και τώρα πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο σε αυτή τη φάση και θα λόγω λόγο στο Χεύμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρα και εγώ θα ήθελα ασφαλώς να ευχαριστήσω την ε, κυρία Γκαρσία Περές για την εξαιρετική της έκθεση ό,τι αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Ευρωπαϊκής ΚΟΑ. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός σύγκλησης μεταξύ της έκθεσης και της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά κυρίως τα βασικά στοιχεία της πρότασης να πω ότι με ικανοποιεί ότι η ανάγκη για τη δημιουργία ενός προτύπου για την αγορά έχει γίνει σωστά αντιληπτή ως τμήμα μιας πιο συνολικής προσέγγισης, μια προσέγγιση πιο πολύ βασισμένη στις ανάγκες της αγοράς θα πρέπει να συμπληρώσει τη συμμόρφωση με βασικούς κανόνες για όλους τους φορείς της αγοράς προς το δικό του συμφέρον. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ε, κυρία Πρόεδρε, για να απαντήσω και στον κύριο Ταντά, ο οποίος ε, εξέφρασε κάποιες αμφιβολίες για τους ελέγχους, να πω ότι θεωρούμε ότι οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να γίνονται και βάσει ανάλυσης κινδύνου και να μην ξεχνάμε ότι ήδη ισχύουν τα γενικά πρότυπα για τη θέση σε εμπορία σε ό,τι αφορά ε, προϊόντα που και για τα οποροκυπευτικά. Άρα δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια δυσκολία. Επίσης, να επαναλάβω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι τα πρότυπα marketing αποτελούν, αποτελεί βασικό στοιχείο του ελέγχου ποιότητας και που επηρεάζει και την ποιότητα του προϊόντος. Ξέρω ότι η προσπάθεια να ενοποιηθεί η νομική βάση με οριζόντια προσέγγιση είναι κάτι το οποίο γίνεται θετικά αντιληπτό. Να τονίσω ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση από πλευράς μας να καταργήσουμε τα ήδη υφιστάμενα πρότυπα ε, marketing. Πρόκειται μια, για μια άσκηση εναρμόνισης και όχι αλλαγής των υφιστάμενων προτύπων. Επίσης, σημειώνουμε ότι σε ό,τι αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας η συγγήτρια θεωρεί ότι είναι ισορροπημένη γενικά η προσέγγιση σε ό,τι αφορά την τροπο, τις τροπολογίες για θεσμικά ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εναρμονίσει και την ε, πρόταση αυτή με, την, ε, με τον κανονισμό για την επιτροπολογία. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της πρότησης, η βασική τροπολογία έχει να κάνει με το κατά πόσο η οι όροι ποιότητα θα πρέπει να καλύπτονται από τον ε, κανονισμό για την, ε, ενιαία ποιότητα, για την ποιότητα της ενιαίας αγοράς και όπως εξήγησα βασικά θέλουμε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να προωθήσουν κάποια χαρακτηριστικά ποιότητας των προϊόντων τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αν ε, συγκεντρώσουμε όλους τους, ε, όλες τις υπονομίες ποιότητας σε ένα κανονισμό, θα είναι πιο συνεπής η προσέγγισή μας. Κάποιες επιπρόσθετες ερωτήσεις να απαντήσω τώρα. Σε ποιο βαθμό τα διεθνή πρότυπα θα ίσχυαν εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαβεβαιώσω τον κύριο Ντάντα ότι αυτά τα διεθνή πρότυπα θα ισχύσουν μόνο αν δεν, υπάρχουν, αν δεν υπάρξει τίποτα πέρα από τα γενικά πρότυπα διάθεσης. Δεν είναι εξαίρεση να ισχύσουν τα διεθνή πρότυπα σε πολλά σε πολλούς τομείς, στον κόντεξ, σε ό,τι αφορά το κρασί, εφαρμόζουμε διεθνή πρότυπα. Γιατί να μην το κάνουμε και εδώ, αν δεν έχουμε εμείς κάτι πιο συγκεκριμένο πέρα από τα γενικά πρότυπα marketing. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κίνδυνο που ανέφερε, ότι τα πρότυπά μας ενδεχομένως να είναι αντίθετα με τα ενδεχόμενα εθνικά πρότυπα. Αυτό δεν θέλουμε να συμβεί και θέλουμε να κάνουμε διευκρινήσεις, ό,τι διευκρινήσεις χρειαστεί στο κείμενο. Εφόσον φυσικά συνάδουμε με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία κανόνες αυτοί. Θεωρούμε ότι η πρότασή μας λοιπόν και βλέπω με χαρά ότι και η συγγήτρια σε μεγάλο βαθμό συμφωνεί με την πρότασή μας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ολοκληρωθεί γρήγορα η διαδικασία για τα προκυπευτικά, για την κατάργηση των συγκεκριμένων προτύπων και τις ενδεχόμενες δυσάρεστες καταστάσεις που μπορούν να προκύψουν. Έγινε μια αξιολόγηση της κατάργησης των προτύπων marketing για τα απορροκυβευτικά, η οποία και κατέδειξε ότι δεν θα, υπήρξαν, δεν θα υπήρχουν διαφορές. Και ότι λίγο πολύ τα ίδια πρότυπα ισχύουν και πάλι. Άρα δεν θεωρούμε ότι υπάρχει κάποια ζημιά από την κατάργηση των συγκεκριμένων προτύπων marketing σε ό,τι αφορά τα οποροκυπευτικά. Να θυμάστε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σχετικά πρότυπα που καλύπτουν το 70% των οποροκυπευτικών. Εξακολουθούν να ισχύουν. Και με αυτό θα ήθελα να κλείσω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Βεσλάινεν Βάιντα πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής του Συμβουλίου για τη Γεωργία. Κύριε Βάιντα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που παραβρίσκομαι εδώ σήμερα. Με ενδιαφέρον άκουσα τις διάφορες απόψεις. Το πακέτο ποιότητας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας και στα πλαίσια του Συμβουλίου εργαζόμαστε εντατικά σε ό,τι αφορά τον έλεγχο αυτής της νομικής πράξης. Μετά από συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας, λοιπόν, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, στα πλαίσια και περαιτέρω ομάδων εργασίας, θα εξετάσουμε τις προτάσεις για την νομοθετική πράξη, θα εξετάσουμε και τις διάφορες πτυχές. 19, συγγνώμη, 17 Απριλίου, στις 17 Απριλίου οι σχετικοί αρμόδιοι υπουργοί θα συνεδριάσουν και θα επεξεργαστούν και το πακέτο ποιότητας. Θέσαμε στα κράτη-μέλη δύο ερωτήσεις και τα παρακαλούμε να μας παρουσιάσουν τις θέσεις τους σε ό,τι αφορά τα τοπικά αυτά προϊόντα και τα προϊόντα της γεωργίας και φυσικά θα υπάρχει η δυνατότητα να συζητηθούν και άλλες πτυχές του πακέτου ποιότητας. Θα υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων. Το Συμβούλιο είναι πρόθυμο να συνεργαστεί επικοδομητικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ασφαλώς βεβαίως και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. E Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να καταλήξετε στα απαιτούμενα συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους ε, της Επιτροπής μας ε, που μου έδωσαν τις απόψεις τους. Να ευχαριστήσω όμως ε, και όλους τους άλλους συναδέλφους. Εν γέννη, νομίζω ότι θα είναι εφικτό να καταλήξουμε σε συμφωνία στο Κοινοβούλιο για τα ουσιώδη. Τουλάχιστον με βάση τα όσα άκουσα, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις που θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να διευκρινίσουμε, αλλά νομίζω ότι τα βασικά ζητήματα όπως είναι ο ρόλος των οργανώσεων παραγωγών, τα προϊόντα ορεινής γεωργίας, ε, οι ορισμοί για τα στάδια παραγωγής, νομίζω από αυτόν θα υπάρξει συμφωνία. Και να ξέρετε ότι είμαστε ανοιχτοί αν υπάρχουν κάποια πιο συγκεκριμένα θέματα για τα οποία θέλετε να κάνουμε κάποια μικρή διαφοροποίηση, μπορούμε να το κάνουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Θα έχουμε σύντομα συνάντηση με τους ε, υπεύθυνους ε, για το θέμα και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Λαμβάνοντας υπόψη τις ε, προτάσεις που ακούσαμε. Αλλά επαναλαμβάνω είναι σαφή τα βασικά σημεία και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Δύο πράγματα μόνο θέλω να αναφέρω. Το πρώτο το είπε η κυρία Μαγκίνες. Νομίζω ότι να απαντήσει σε αυτό ε, αρμόδια είναι η Επιτροπή για την ε, σήμανση προέλευσης. Πρόκειται για τον κανονισμό περί πληροφόρησης ε, και ενημέρωσης των καταναλωτών. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση της κυρίας Μαγκίνες. η δική μας επιτροπή έχει αποφανθεί όταν βλέπαμε κατά περίπτωση κάποια πράγματα και θα δούμε και στη συνέχεια τι απάντηση θα δώσει η Κομισιόν. Και κάτι ακόμη. σε σχέση με προαιρετικού αποκλειστικούς όρους. Αν στόχος μας είναι να ενισχύσουμε το σύστημα ποιότητας, και υπάρχει και γι' αυτό το λόγο κανονισμός ποιότητας, που έχουμε δύο επίπεδα. Έχουμε προστατευόμενε ονομασίε προέλευση, γραφικέ ενδείξει και εγκυμένα ειδικά παραδοσιακά προϊόντα, που είναι ο καλύτερο δυνατό τρόπο να προστατεύσουμε την ποιότητα των προϊόντων μα. Και έπειτα έχουμε κάποιε προαιρετικέ ενδείξει, που είναι οι προϊόντα ορεινή γεωργία κτλ. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Ένα αυτό και άλλο τα υπόλοιπα προϊόντα, που το μόνο κοινό που έχουν είναι ότι είναι προαιρετικά. Γιατί ουσιαστικά είναι να λέμε στους καταναλωτές ότι το προϊόν ε, είναι σύμφωνο με μια συγκεκριμένη μέθοδο γεωργίας εκτινοτροφίας. Όταν μιλάμε για την ε, πίεση ψυχρό του ελαιολάδου και κάτι άλλο σχετικά. Τι σχέση έχει αυτό με πραγματική ονομασία προέλευση ή γεωγραφική ένδειξη, οι οποίε είναι προστατευόμενε και όπου εκεί πραγματικά αναφέρονται οι προποθέσει που πρέπει να πληρούνται για να έχει αυτή την ονομασία ή ένδειξη ποιότητα στο εν λόγω προϊόν κάθε φορά. Άρα το μόνο κοινό σημείο που έχουν αυτοί οι όροι με τα υπόλοιπα ε, συστήματα ποιότητα είναι ότι είναι προαιρετικά όλα αυτά. Δεν νομίζω όμω ότι αυτό αποτελεί λόγο επαρκεί για να το συμπεριλάβουμε και να φέρεται στα πρότυπα ε, της εμπορίας της κοινή οργάνωσης αγοράς. Θέλουμε ένα ισχυρό σύστημα. Το είπα και το ξαναείπα. Θέλουμε επίσης ένα σύστημα ποιότητας που να προστατεύονται αυτά τα προϊόντα, τα ποιοτικά. Αν αναφέρουμε λοιπόν αυτές τις προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας, ουσιαστικά αυτό αποδυναμώνει το σύστημα ποιότητας. Καταλαβαίνω ότι στα πρότυπα εμπορία ε, τη Ενιασκόας θα πρέπει να ε, τα εντάξουμε αυτά. Ολοκληρώνοντα, θέλω να πω ότι είμαι ε, στη διάθεση των συναδέλφων από την Επιτροπή μα. Σίγουρα θα χρειαστεί η πρόταση αυτή κάποιες βελτιώσεις για να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις και νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για να έχουμε μια ισχυρή θέση έναντι και των διαπραγματεύσεων που επαναλαμβάνω και με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο νομίζω θα έρθω σε αίσιο πέρας. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η Ράση. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους ε, ομιλητές της Επιτροπής μας και τους προσώπους της Κομισιόν και την Ειδική Επιτροπή, τον Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής κ. Βάιντα. Το τελευταίο σημείο για σήμερα είναι τροποποίηση του κανονισμού 1290 του Συμβουλίου και κατάσταση κανονισμών 165 και 78. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για την ευθυγράμμιση του κανονισμού με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ο εισηγητής θα μας παρουσιάσει τις τροπολογίες που έχει προετοιμάσει. Ευχαριστώ τον Διευθυντή Λόγκο που είναι εδώ από την Επιτροπή και θα δώσω το λόγο στον Λαβία θυμίζοντας ότι η προθεσμία της κατάθεσης τροπολογιών είναι η 3η Μαρτίου, ήτανε 3η Μαρτίου 12η ε, μεσημβρινή στις 25 Μαΐου θα γίνει ψηφοφορία. Τζοβάνι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας ήταν απαραίτητη αυτή η προσπάθεια ευθυγράμμισης και του κανονισμού 1290 του 05 με τις ισχύουσες συνθήκες πλέον και σχετικά με τις προερχόμενες αρμοδιότητες για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε αυτά τα οποία προεβλέπονται σε αρχικό επίπεδο από τον κανονισμό. Μετά την εξέταση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί τη βάση των, των συγκεκριμένων δύο κατηγοριών, είδαμε ε, ποια είναι τα πλαίσια στα οποία οι προερχόμενες αυτές ε, πράξεις ε, είναι αποδεκτές και σε σχέση με τις εκτελεστικές πράξεις. Στην ουσία ακολουθήσαμε μια γραμμή συμβατή με αυτά τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη κάνει γενικότερα με το θέμα της ευθυγράμμισης για τους υπόλοιπους κανονισμούς. Παρουσιάσαμε λοιπόν κάποιες προτάσεις λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που έχουν κάνει ορισμένα εθνικά κοινοβούλια για ορισμένες τροπολογίες που αφορούν τις ε, ε, προϋποθέσεις της, ε, της εκχώρησης αυτής της αρμοδιότητας, τη διάρκεια, την παράταση, της, την επιτροπολογία κτλ. Παρουσιάσαμε τις τροπολογίες αυτές σύμφωνα πάντα με την κοινή προσπάθεια που κάνουμε για τους πρακτικούς τρόπους προσφυγής στις προερχόμενες αυτές ε, πράξεις σύμφωνα με την απόφαση της 3ης Μαρτίου 2011 και σύμφωνα με τον κοινό κανονισμό του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Ο τελευταίος αυτός κανονισμός καθορίζει τους κανόνες, τους βασικούς με τους τρόπους ελέγχου από πλευράς των κρατών μελών των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων οι οποίες δίδονται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιες από τις τροπολογίες τις οποίες παρουσιάσαμε αφορούν το θέμα της απλοποίησης. Ιδιαίτερα σκοπεύαμε να απλουστεύσουμε την τυπολογία των δαπανών στα πλαίσια του ΦΕΟΓΚΑ, την διαδικασία ανάκτησης σε επίπεδο διοικητικής διαδικασίας και στη μείωση των διοικητικών δαπανών εις βάρος των κρατών μελών. Προτείναμε επίσης και άλλη μία τροπολογία, την σχετική με το άρθρο 29 του κανονισμού 1290 Προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε τους όρους για την ανάπτυξη της υπαίθρου σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο. Όπως όλοι γνωρίζετε σήμερα, τα κράτη-μέλη τα οποία αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους για την ανάπτυξη της υπαίθρου σε περιφερειακό επίπεδο, βλέπουν την ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτού σε σχέση με τα μεμονωμένα λειτουργικά προγράμματα χωρίς να προβλέπεται ένα ευρύτερο πλαίσιο εθνικό Γι' αυτό ακριβώς το λόγο προτείναμε μια συγκεκριμένη τροπολογία η οποία προβλέπει μπορεί να προβλέψει μια εθνική αντιστάθμιση έτσι ώστε να διατηρηθεί όσο περισσότερο γίνεται το ανώτατο όριο το οποίο δίδεται στα διάφορα ε, Ευχαριστώ Τζοβάνι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος συνάδελφος που παίρνει το λόγο, αλλιώς θα δώσω αμέσως ε, το λόγο στον, επίτρο... στον εκπρόσωπο Λόγκο, τον Διευθυντή κύριο Λόγκο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου και εμένα να ευχαριστήσω τον κύριο Λαβία για το σχέδιο εκθεσής του, το οποίο παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. metà, certamente per la metà degli emendamenti eh, proposti. Και θα συμφωνήσουμε με τις περισσότερες από τις τροπολογίες τις οποίες προτείνει. Θα θέλαμε να εκφραστούμε θετικά για τις τροπολογίες 1, 2, 8, 9 και 10. Στο βαθμό που οι τροπολογίες αυτές, όπως το είπε ήδη ο κύριος Λαβιάχ, είναι συνεκτικές με την κοινή προσπάθεια την οποία κάνουμε και είναι αποδεκτές συνεπώς για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέραν αυτού θα ήθελα να προκαταλάβω όμως το συγκεκριμένο θέμα να πω για την κοινή προσπάθεια η οποία αφήνει σε εκκρεμότητα την δυνατότητα που υπάρχει περιορισμού χρονικού της απόδοσης εξουσιών ή μάλλον αρμοδιοτήτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως προτείνεται στην τροπολογία υπαρίθμε 7. Πιο συγκεκριμένα και σχετικά με τις τροπολογίες 3 και 4 διαπιστώνουμε ότι με έμεσο τρόπο ζητείται, στοχεύεται μάλλον η κατάργηση της αναφοράς στην απόφαση του Συμβουλίου. Αυτό σημαίνει υπάρχει, ότι υπάρχει μια αλλαγή της διαδικασίας στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχία όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 του κανονισμού 73 του 2009 αυτό είναι ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Νομίζω ότι σε μια άλλη συζήτηση που είχατε κάνει στην Επιτροπή σας το είχατε έχει. Είναι σαφές ότι υπάρχει σύνδεσμος και με το θέμα της αλλαγής της διαδικασίας σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές γύρω από τον κανονισμό 73 και 90. Από πλευρά μα εμείς θεωρούμε και είχαμε ήδη τη δυνατότητα να εκφραστούμε περί αυτού ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να δράσει επί τη βάση του άρθρου 43.3 της Συνθήκης για τη Δημοσιονομική Πειθαρχία. Σχετικά τώρα με την ποσόστοση τη δημοσιονομική, τη λεγόμενη ρύθμιση στο κείμενο, περιοριζόμαστε στην εφαρμογή των άμεσων πληρωμών, δηλαδή στο επίπεδο βοηθειών, επιδοτήσεων οι οποίες έχουν δοθεί. Αυτό είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση 43-3 και αυτό νομίζω εξηγείται πλήρως από το κείμενο της Νέας Συνθήκης. Επί τη βάση της νέας αυτής συνθήκης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει μια σαφέστατη διάκριση και το έχει ήδη πει αυτό η ΣΥΙΤΙΣ ανάμεσα στους διαφορετικούς εφαρμόσιμους κανόνες, στα διαφορετικά εφαρμόσιμα άρθρα. Συνεπώς εμείς πιστεύουμε ότι ο καθορισμός των συγκεκριμένων αυτών ρυθμίσεων σε σχέση με την ποσόστοση που θα πρέπει να εφαρμοστεί στις επιδοτήσεις τις οποίες παίρνουν οι γεωργοί και στα πλαίσια των δημοσιονομικών προβλέψεων από τη μία και σε σχέση με τα στοιχεία που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τύχει η λήψη απόφασης. Να επανέλθω τώρα με μια άλλη πλευρά η οποία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον μια άλλη διάσταση αν θέλετε του συγκεκριμένου θέματος. Πράγματι το Συμβούλιο δεν δρά σαν νομοθέτη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Περιορίζεται όμως την αντίδραση απλά χωρίς καμία δυνατότητα κίνησης, κανένα περιθώριο κίνησης στις δημοσιονομικές συνθήκες οι οποίες καταρχάς αποφασίζονται από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή, δηλαδή από εσά. Δίνε πως θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η αποδοχή μιας νομοθετικής πράξης μέσα σε τρεις μόνο μήνες, γιατί αυτό προβλέπεται για την εφαρμογή ακριβώς αυτής της δημοσιονομικής ρύθμισης, είναι κάτι το όχι πολύ ρεαλιστικό. Ω εκ τούτου το να συνδεθεί το Κοινοβούλιο με τη διαδικασία αυτή σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παραμείνει μόνη να λάβει αποφάσεις σχετικά με τους όρους εφαρμογής της δημοσιονομικής αυτής ρύθμισης. Αντίθετα τώρα σχετικά με την τροπολογία 5. Η τροπολογία 5 προβλέπει την υιοθέτηση μέτρων οι οποίες, ε, τα οποία έχουν υποβληθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να καταστούν ε, οι προτάσεις στις συμβατές με το ανώτατο όριο το προβλεπόμενο από το άρθρο 12 παράγραφος 3. Νομίζω ότι αυτά ανήκουν όπως και να έχουν τα πράγματα στην εφαρμογή του άρθρου 43 παράγραφος 2 της συνθήκης. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η δυνατότητα αποκλειστικής αποδοχής από πλευράς του Συμβουλίου μόνον μπορεί να υπάρξει στην περίπτωση κατά την οποία πρόκειται για ένα θέμα σχετικό με τον καθορισμό του ύψους της επιδότησης. Για το τελευταίο σημείο. Ε, πρόκειται για μια τροπολογία, η εξι η οποία είναι επί της ουσίας και όχι επί της διαδικασίας. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτρόπης είναι μια πρόταση η οποία έχει σαν μοναδικό στόχο το να εμείνουμε στην απλή προσαρμογή στη συνθήκη και ως εκ τούτου δεν θέλουμε να προχωρήσουμε πέραν αυτού και γι' αυτό εμένουμε στην διάσταση αυτή, την προσαρμοστική θα έλεγα προς τη συνθήκη και δεν σκοπεύουμε να προχωρήσουμε πέραν αυτού. Θα ήθελα συμπερασματικά να αναφερθώ στο πρόβλημα της διάρκειας των κατεξουσιοδότηση πράξεων που εκχωρούνται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο περιορισμός του ο χρονικός την πενταετία μόνον μπορεί να δημιουργήσει μια σειρά από βασικά προβλήματα διότι διατρέχουμε τον κίνδυνο να δημιουργηθεί μια κατάσταση ασυνέχειας στα πλαίσια της εφαρμογής του συγκεκριμένου κανονισμού, κάτι το οποίο θα δημιουργούσε σημαντικότατα προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να συστήσω αυτό το οποίο είναι κατά τα άλλα εφικτό, να προσανατολιστούμε δηλαδή σε μία επιλογή εκχώρησης αρμοδιότητας χωρίς χρονικό περιορισμό, όπως ακριβώς το κάνει το Συμβούλιο, χωρίς να υπάρχει δηλαδή χρονικός περιορισμός. Πάντως το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν μια ελεγκτική αρμοδιότητα της ε, κατεχώρηση νομοθετικής αυτής ρύθμισης της Ευρωπαϊκής Επίτροπης που παρέχει όλες τις απαιτούμενες εγγυήσει για τη συνέχεια της διάρκειας αυτής της πράξης. Ευχαριστώ τον Διευθυντή κύριο Λόγκο και θα δώσω το λόγο πάντα στον κύριο Λαβία. Εδώ θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω <clears throat> την αναφορά στο άρθρο 43 Το άρθρο 43 ακριβώς είναι αυτό το οποίο δημιουργεί τα σημαντικότατα προβλήματα γιατί αποκλείει το Κοινοβούλιο από τις επιλογές που λαμβάνονται και είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ στο συγκεκριμένο αυτό κείμενο περί της χρηματοδότησης ή στα πλαίσια των υπολείπων πράξεων των προσαρμοστικών να μπορέσουμε να βρούμε μια συμφωνία πάνω σε αυτό το άρθρο το οποίο όπως είπα αποκλείει κάθε ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχει συγκεκριμένο ρόλο και είναι διατεθειμένο να επιδιώξει να αναλάβει τις αρμοδιότητες τις οποίες του αποδίδει η συνθήκη ιδιαίτερα στον δημοσιονομικό τομέα. Γιατί επαναλαμβάνω, στον δημοσιονομικό τομέα η ίδια η συνθήκη της Λισαβόνας ξεκαθαρίζει σαφέστατα το τμήμα ε, για το οποίο είναι υπεύθυνο το Κοινοβούλιο. Και ξαναγυρνάω στον εισηγητή, τον κύριο Λαβία. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθύντη κύριο Λόγκο, ο οποίος μας παρουσίασε τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχω να πω τίποτα, δεν έχω να σχολιάσω πάνω στις τροπολογίες για τις οποίες υπάρχει ήδη συμφωνία. Τροπολογίες οι οποίες μπορούν να θεωρούνται πλέον δεκτές και μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι όμως σαφές ότι στα υπόλοιπα θέματα υπάρχει θα έλεγα μια διαφορετική άποψη. Η έκθεση δεν είναι κάτι το τεχνικό απλά, είναι κάτι το οποίο υπογραμμίζει και τον πολιτικό ρόλο του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο θέλει να εμπλακεί στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων και να μην παραμένει μακριά, μακρινός μάρτυρας της κατάστασης. Απλά για το θέμα των επιστροφών. Και σχετικά με την τελευταία τροπολογία, είναι αλήθεια ότι είναι μια τροπολογία, όπως είπε ο κύριος Λόγκο, ουσίας. Αυτή τη στιγμή εμείς υιοθετήσουμε μια νέα διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει την δυνατότητα να την κρίνει, να την εγκρίνει. Και είναι λοιπόν θεμητή η προσδοκία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της δικής μας Επιτροπής συγκεκριμένη περίπτωση, να κάνει κάποιες πιθανές αλλαγές τροποποιήσεις στο κείμενο του κανονισμού. Κατανοώ βέβαια ότι εδώ άπτεται το θέμα της ουσίας και επί της ουσίας δεν αναφέρθηκε ο, ο κύριος Διευθυντής, αλλά από την άλλη είναι σαφές ότι έχουμε να κάνουμε με μια βασική γραμμή στην οποία θα εμείνει το Κοινοβούλιο και θα προτείνει ε, προς ψηφοφορία την άποψή του, η οποία είναι κατευθυντήρια γραμμή και για το Συμβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σαφές ότι θα επανέλθουμε στο εσωτερικό της Επιτροπής μας για το θέμα ε, θα δούμε αν στα πλαίσια των προθεσμιών τις οποίες υπέδειξε ο πρόεδρος Δεκάστρο θα έρθουν και άλλες ε, τροπολογίες, θα μεσολαβήσουν και άλλες τροπολογίες. Σας ευχαριστώ όλους. Ε, τέλος της συνεδρίασης. Σας θυμίζω ότι αύριο στις 9 έχουμε τους συντονιστές και στις 9 και 30 έχουμε τη συνεδρίαση την κανονική.